Καλησπέρα σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, θα θέλαμε οι διερμηνείς να ενημερώσουμε ότι βρισκόμαστε στην 35η μέρα τις ε, διαμαρτυρίες μας ε, για τις απαράδεκτες συνθήκες που έχουν επιβληθεί οι συνθήκες εργασίας στους διερμηνείς του Κοινοβουλίου. Λυπούμεθα, αλλά θα θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν θα υπάρξουν υπερβάσεις ωραρίου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Βλέπω ότι έχετε υιοθετήσει την ιδέα να κάνουμε μια απογευματινή συνεδρίαση. Όπως ακούσατε και από το μήνυμα, υπάρχει μια δράση των διερμηνέων. Πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Ο πρόεδρος λέει θέλω να ζητήσω από του διερμηνείς να μας παρουσιάσουν τη γλωσσούς. Ακούσατε ήδη το μήνυμα από τους διερμηνείς. Well, and thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Το πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερησίας διάταξης. Ελπίζω όλοι να έχετε δει ποιο θα είναι το πρόγραμμα της σημερινής σας συνεδρίασης. Υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι, σας ευχαριστώ. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερησία διάταξη. Δεύτερο σημείο έγκριση των ε, πρακτικών των συνεδριάσεων 16-17 Μαΐου 2018. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Επομένως, αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης, θα θεωρηθούν εγκριθέντα. Να ξεκινήσουμε, λοιπόν, με το πρώτο ουσιαστικό σημείο του προγραμματός μας. Μέχρι τις 4 και 10 έχουμε δηλαδή 40 λεπτά για την έκθεση σχετικά με τις υποδομές ευρωζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας παρουσίαση από την κυρία Ηλιάνα Ιβάνοβα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Θα ήθελα να την παρουσιάσω Να σας υπενθυμίσω ότι η κυρία Ιβάνοβα είναι επικεφαλής του τμήματος 2 στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο υπεύθυνη για τους ελέγχους στον τομέα επενδύσεων για τη συνοχή, την ανάπτυξη και την συμπερίληψη. Έχουμε 40 λεπτά, όπως σας είπα για το θέμα αυτό. Θα ήθελα επομένως να προτείνω η κυρία Ιβάνοβα να παρουσιάσει μέσα σε 10 λεπτά το θέμα, κατόπιν να πάρουν το λόγο οι συντονιστές, οι αντικαταστάτες των συντονιστών, για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους εντός 2 λεπτών και όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέλη έχουν ένα λεπτό στη διάθεσή τους. Στη συνέχεια θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Ιβάνοβα να απαντήσει ή να σχολιάσει Και στη συνέχεια ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα σε αυτή την Επιτροπή. Συνήθως ε, παρουσιάζομαι τις περισσότερες εκθέσεις στην Επιτροπή Κοντ. Βλέπω και κάποιους ε, πρώην συναδέλφους από εκεί εδώ σήμερα. Για μένα είναι πρώτη φορά βέβαια στην Επιτροπή Βιομηχανίας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την πρόσκληση για να σας παρουσιάσω αυτό το πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα, την ε, ευρυζωνική κάλυψη. Είναι κάτι που θα μπορούσα να φανταστώ ότι είναι μέρος της ζωής όλων μας. Όλοι χρησιμοποιούμε υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και για να έχουμε πρόσβαση στο διαδίκτυο χρειαζόμαστε καλή ευρυζωνική κάλυψη. Έτσι λοιπόν ο τίτλος τη Ειδική Έκθεση που θα σα παρουσιάσω είναι ευρυζωνική σύνδεση στα κρατη παρά την πρόοδο δεν θα πετύχουμε όλου τους στόχους της Ευρώπη το 2020. Εδώ ο όρος ε, χρησιμεύει για να ε, περιγράψουμε τις ε, πιο υψηλές ταχύτητες στο ίντερνετ. Οι καλές συνδέσεις στο ίντερνετ είναι σημαντικές όχι μόνο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να μην είναι παγκοσμίω, αλλά και για την πρόθεση της κοινωνικής ένταξης. Τώρα, ποιο είναι το σημείο αφετηρίας στη Στρατηγική Ευρώπη 2020. Έχουμε το ψηφιακό θεματολόγιο με τρεις κυρίους στόχους το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τους στόχους ε, για τις ευρυζωνικές ε, συνδέσεις ε, που σχετίζονται με τη βασική ευρυζωνική σύνδεση, δηλαδή μέχρι 30 MB ανά δευτερόλεπτο, για να διασφαλίσει ότι μέχρι το 2013 όλοι οι πολίτες θα έχουν να έχουν σύνδεση. Μέχρι το 2020, ε, ως το δεύτερο στόχος, ήταν να έχουν γρήγορη βριζονική, δηλαδή ταχύτητα μεταξύ 30 και 100. Και ο τρίτος στόχος ε, είναι μέχρι το 2020 και πάλι να διασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 50% των οικοκυριών θα έχουν ε, πρόσβαση σε πολύ γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση, δηλαδή ταχύτητα πάνω από 100 ε, ΜΜ. δηλαδή μέχρι το 30 είναι η βασική, από 30 μέχρι 100 η γρήγορη και η πάρα πολύ γρήγορη, πάνω από 100 MB ένα δευτερόλεπτο. Και για να υποστηρίξουμε τους στόχους αυτό, έχουμε μια σειρά μέτρων κανονιστικών και μέτρων πολιτικής. Ποια είναι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι περίπου 15 δισεκατομμύρια για την περίοδο 14-2020 με μία πηγή πηγών χρηματοδότησης. Έχουμε επιχορηγήσεις από τον Ευρωπαϊκό Υπολογισμό. Έχουμε πόντα 6 δισεκατομμύρια σε δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης έχουμε τα project του ΕΦΣΙ, Έχουμε λοιπόν μία μεγάλη ποικιλία χρηματοδότησης. Τώρα, που επικεντρώσαμε τον έλεγχό μας. Προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα των δράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών για την επίτευξη αυτών των τριών στόχων μέχρι το 2020 και θέλαμε να αξιολογήσουμε αν τα κράτη-μέλη πρόκειται να πετύχουν τους στόχους αυτούς και αν η Κομισιόν ε, παρακολουθεί αυτά τα επιτεύγματα. Επίσης, αν τα κράτη-μέλη έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων και βεβαίως αν είχαν αποτελεσματικά εφαρμόσει αυτές τις στρατηγικές, δηλαδή όχι μόνο να τις έχουν σχεδιάσει αλλά και να τις έχουν εφαρμόσει. Ο έλεγχος καλύπτει την περίοδο 2014-2020 και την περίοδο 2007-2013 και όλες τις πηγές χρηματοδότησης και την στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως σας ανέφερα. Βλέπετε στη διαφάνεια, επισκεφτήκαμε πέντε κράτη-μέλη, Ιρλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ιταλία όπου είχαμε συζητήσεις με μια σειρά άλλων ενδιαφερομένων μερών σημαντικών. Στην επόμενη διαφάνεια δεν ξέρω αν ε, είναι ιδιαίτερα εύληπτη, δεν θα τη σχολιάσω ιδιαίτερα, αλλά βλέπετε μια απεικόνηση της κατάστασης ε, της ε, γρήγορη ευρυζωνικής σύνδεσης το 2016 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη ε, από 30 μέχρι 100 βλέπετε ότι οι πιο πράσινες περιοχές είναι που είναι πιθανότερο να επιτευχθούν οι στόχοι και με το πιο ανοιχτό πράσινο είναι που είναι πιο χαμηλό το ποσοστό. Βλέπετε λοιπόν από το χάρτη ότι σαφέστατα δεν θα έχουμε επιτυχία μέχρι το 2020. Πιθανότατα. Το γενικό μας συμπέρασμα από το συνολικό έλεγχο είναι ότι κάποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί, ο βασικός στόχος της ε, βασικής κάλυψης, δηλαδή μέχρι 100 MB ένα δευτερόλεπτο. Βασικά όλα τα κράτη-μέλη το πέτυχαν αυτό μέχρι το 2016. Αν ε, και η προθεσμία στη στρατηγική ήταν 2013, αυτός ήταν ο στρατηγικός στόχος, αλλά μέχρι το 2016 πάνω κάτω όλοι είχαν διασφαλίσει ότι υπάρχει κάλυψη για βασική ευρυζωνική σύνδεση. Όμως, ε, τους υπόλοιπους δύο στόχους, τη γρήγορη και την ε, πάρα πολύ γρήγορη, δεν το χάρτη για τη γρήγορη, για την υπερβολικά γρήγορη κατάσταση είναι ακόμη λιγότερο υποσχόμενη. Και οι αγροτικές περιοχές, ε, ε, η Ήπεθρος είναι πιο προβληματική σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Μέχρι τα μέσα του 2017, 14 κράτη-μέλη είχαν κάλυψη στην Ήπεθρο λιγότερο από 15% και για τον ε, τρίτο στόχο μόνο το 15% των οικοκυριών είχε ε, ουσιαστικά αυτή την ε, ταχύτητα στη σύνδεση. Έτσι λοιπόν, 15% ε, είχαμε επιτυχία, έναντι του στόχου 50%. Παρόλα αυτά τα προβλήματα, αν τα σχέδια των κρατών μελών εφαρμοστούν όπως σκοπεύεται, τρία από αυτά τα πέντε κρατημέλη που επισκεφτήκαμε μπορεί να είναι σε μια καλή θέση να πετύχουν τους στόχους της Κομισιόν για το 2025. Ότι δηλαδή όλα τα νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ιδιαίτερα γρήγορη σύνδεση. Η υποστήριξη της Κομισιόν που δόθηκε στα κρατημέλη αξιολογήθηκε επίσης από εμά και ενώ αξιολογήθηκε θετικά από αυτούς, εμείς βρήκαμε ότι δεν υπήρχε συντονισμός ε, μεταξύ των διαφορετικών διευθύνσεων της Κομισιόν. Τώρα, κάποιες από τις αδυναμίες που ανακαλύψαμε στις στρατηγικές. Παρατηρήσαμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν αναπτύξει τέτοιες στρατηγικές ε, ευρυζωνική σύνδεση, αλλά σε αυτά που εξετάσαμε βρήκαμε κάποιες ελλείψεις, ε, κάποια κράτη-μέλη είχαν καθυστερήσει στο να ολοκληρώσουν τι στρατηγικέ. Μερικές φορές οι στόχοι δεν ήταν πάντοτε συνεκτικοί με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Κανένα από τα κρατημέλη που επισκεφθήκαμε μάλιστα δεν είχε θέσει ως στόχο τον ε, τρίτο που σας ανέφερα στην αρχή. Δηλαδή την πρόσληψη πάρα πολύ γρήγορης ε, ευρυζωνικής σύνδεσης. Αυτό δεν ήταν μέρος των στρατηγικών που αναλύσαμε. Επιπρόσθετα, δεν είχαν αντιμετωπίσει όλα τα κρατημέλη τις προκλήσεις ε, που σχετίζονται με τις ε, υποδομές, ε, δηλαδή με τις τηλεφωνικές επιδομές, με τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να υπάρχουν στις ταχύτητες των συνδέσεων. Ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορες επιλογές υποδομής όπως ε, το χάρη, το παραδοσιακό ε, μοντέλο είναι τα δίκτυα χαλκού, αλλά ε, έχουμε βέβαια και άλλες τεχνολογίες, όπως ασύρματες τεχνολογίες, υπάρχουν διάφορες λύσεις, αλλά και διάφορες επιπλοκές ανάλογα με τις επιλογές των κρατών μελών. Τώρα, κάτι που ήταν ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ήταν διάφορους περιοριστικούς παράγοντες στην ε, πρόοδο για την επίτευξη των στόχων. Ο πρώτος περιοριστικός παράγοντας ε, πάντοτε σχετίζεται με τη χρηματοδότηση. Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν από την Κομισιόν, το ποσό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του 2020 εκτιμόταν με στα 250 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η εκτίμηση του 2013 και η EIB εκτίμησε ότι το ίμιση του κόστους αφορούν την ύπεθρο που το 20% του πληθυσμού κατοικεί. Και είδαμε ότι η χρηματοδότηση στις αγροτικές περιοχές δεν είχε δοθεί επαρκώς σε τρία από τα πέντε κρατημέλη. Εξετάσαμε την κατάσταση και ανακαλύψαμε ότι ένα μεγάλο project της Τράπεζας Επενδύσεων στηρίχθηκε από το ΕΦΣΥ αλλά δεν επικεντρώθηκε στην πραγματικότητα σε αυτές τις περιοχές ε, όπου χρειάζεται περισσότερο η στηρίξη από το δημόσιο τομέα. Ένας άλλος ε, παράγοντας που εντοπίσαμε ήταν ε, το ανταγωνιστικό και το νομικό περιβάλλον που έθετε πρόβλημα σε δύο κράτη-μέλη, Ιρλανδία και Γερμανία. Εκεί ανακαλύψαμε κάποια προβληματάκια και τέλος η πτυχή που σχετίζεται με τον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των διαφορών πηγών χρηματοδότησης ε, και των ε, μακρών περιόδων. Είδαμε ότι το κατάλληλο επίπεδο συντονισμού εσφάλισε οικονομίες κλίμακας ε, σε τρια κρατημέλη, όμως σε δύο από αυτά, λόγω διάφορων θεμάτων, επειδή υπήρχε παραδείγματο χάρη δύσκολο συντονισμό μεταξύ των προγραμματικών περιόδων, αυτό το πρόβλημα του συντονισμού αποτέλεσε έναν παράγοντα αναστολή τη πρόοδου. Τώρα, φυσικά όπως σε κάθε έκθεση έχουμε και εδώ συστάσει βάσει των πορισμάτων κάνουμε 8 συστάσεις στην Κομισιόν. Στρατηγικό σχεδιασμός, ρυθμιστικό κανονιστικό περιβάλλον, πρόθεση του ανταγωνισμού και δηλαδή να συστάθουν στα κράτη-μέλη να αναπτύξουν αναθεωρημένα σχέδια προκειμένου να πετύχουν τους νέους στόχους. Επίσης, συστήνουμε όλα τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν τις εντολές των εθνικών ρυθμιστικών τους αρχών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο στον τομέα του ανταγωνισμού και του και του νομικού και σε κάποια διαφάνειες σας παρουσίασα περί τίνος πρόκειται. Αλλά φυσικά είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Well, thank you very much, madam, for your introductory remarks. Maybe uh, Mr. Romuald Kaimbada, who came alongside with you, could add some remarks. Would you like to add something to the presentation? No. Okay. So, oh, that's great. The first one to get possibility to express her idea. Θα μιλήσει. Είναι ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ. Okay. Bonnie. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμη κατά την άποψή μας, όχι μόνο για να ε, δούμε πώς αξιολογείται γενικά την ε, κατάσταση, αλλά και γιατί ε, όσο συζητούμε για τα θέματα αυτά και μάλιστα αύριο θα ψηφίσουμε και για τον κώδικα ηλεκτρονικού χώρου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ε, βεβαίω το ευρωζωνικό σύστημα αποτελεί τη βάση. Λοιπόν, ζητήσατε, ρωτήσατε να μάθετε από τα κράτη-μέλη για το ψηφιακό περιβάλλον και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν ε, να επιτευχθούν οι παλιοί στόχοι με την ε, επόμενη τα το 5G, γιατί σε ορισμένες χώρες δεν είναι πολύ σαφής η διαδικασία ολοκλήρωσης των προηγουμένων στόχων και της ταυτόχρονης εκκίνηση των νέων στόχων που θα εστιάζονται στο 5G. Δεύτερη ερώτηση, σε σχέση με τις εθνικές στρατηγικές. γιατί είδαμε τις απαιτήσει που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Από την άλλη πλευρά, οι απαιτήσει για 5G λένε ότι το ότι το 17, τέλη 17, αρχές 18 θα έπρεπε να ε, ε, υπάρχει το νέο ευρυζωνικό εθνικό σχέδιο. ποιες είναι οι δυνατότητες να ολοκληρωθούν, να ολοκληρωθούν ε, οι παλιές αυτές διαδικασίες ενώ ταυτόχρονα προετοιμαζόμαστε για τις νέες προκλήσεις. Ε, εξ όσων γνωρίζετε, τι συμβαίνει και ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Τρίτον, είπατε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και το γνωρίζουμε και εμείς φυσικά σχετικά με την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και την ποιότητα ε, του ε, ίντερνετ ε, στις περιοχές της υπαίθρου. Βεβαίως το ένα πρόβλημα σχετίζεται με τον πληθυσμό αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι ο μόνος λόγος. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή Κατά την άποψή σας ε, υπάρχουν και άλλοι λόγοι και ποιοι είναι αυτοί. Επίσης, όταν μιλάμε για αριθμιστικό περιβάλλον, δεν ε, αναφερθήκατε στο φάσμα και την κατανομή του φάσματος. Ε, υπάρχει κάποια σχέση με την κατανομή του φάσματος στις χώρες που αναφέρατε ή όχι, γιατί οι στόχοι 13-15 ε, και 1500 ε, MB ανά δευτερόλεπτο είναι οπωσδήποτε προκλήσεις οι οποίες σχετίζονται και με αυτές που ανέφερα μόλις προηγουμένως. Ευχαριστώ. Ξεπεράσατε, λέει ο Πρόεδρος, τον χρόνο σας, αλλά εν πάση περιπτώσει η κυρία Βεϊκούνεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την ε, ε, εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί το θέμα ε, τούτο είναι ιδιαίτερο σημαντικό για ολόκληρη την Ευρώπη. Το θέμα των των επικοινωνιών και των διασυνδέσεων είναι πολύ σημαντικές. Αξιολογήσατε πέντε διαφορετικές χώρες. Βρήκατε καλά παραδείγματα όμως. Δηλαδή Υπάρχουν καλά διδάγματα, υπάρχουν κάποια θέματα ε, στα οποία διαπιστώσατε επιτυχία, σημεία τα οποία θα μπορούσαν να μοιραστούν με άλλες χώρες. Επίσης, ε, ο ρόλος ε, του στρατηγικού σχεδιασμού και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος τα αναφέρατε αυτά. Υπάρχουν όμως και άλλα εργαλεία βρήκατε κάποια, διαπιστώσατε την ύπαρξη προβλημάτων ας πούμε οι περιοχές που ανέφερε και ο κύριος Μπόνη προηγουμένως όπου δεν υπάρχει καλή κάλυψη ε, ποια είναι τα επιπλέον εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βρεθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση. Ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις σας. Επόμενος ομιλητής. Υπάρχει εκπρόσωπος ε, της ομάδας Άλντε. Όχι. Πράσινοι έχουν εκπρόσωπο, όχι. Ο αγαπητός συνάδελφος ο Τιγκούε θέλει το λόγο, όχι. Άλλα σχόλια. FDD, NF. Other participants. Κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες μήπως. Ε, αλλά εγώ να πάρω το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Γιατί και εγώ συμμετέχω ενεργά. Ερώτηση λοιπόν είδαμε έναν χάρτη πολύ στον, στην παρουσίασή σας. Είναι ενδιαφέρον ότι εκεί που υπάρχει πυκνότητα πληθυσμού ε, έχει υπάρξει υποδομή για ευρυζωνικότητα στις μεγάλες πόλεις κλπ. Αλλά είδα και στην Νότια Ιταλία κάτι αντίστοιχο. Γιατί Μιλάμε για ε, καθαρά περιοχές της Υπέθρου, στον Πάρι ας πούμε. Παρά τα πολλά χρήματα τα οποία έχουν δοθεί στην ε, περιφέρεια αυτή. Τι γίνεται, τι έχει συμβεί εκεί. Ενώ είδαμε ότι οι αντίστοιχε περιοχές της Γαλλίας ας πούμε έχουν ένα πολύ απαλό πράσινο χρώμα. Άρα, άρα δεν είναι πολύ αποτελεσματική η παρουσία της ευρωζωνικότητας και είδαμε ότι υπάρχουν πολλές ελλείψεις σε μεγάλες ευρείες περιοχές της Γαλλίας όσον αφορά αυτό το ταχύ ίντερνετ. Την απάντησή σας κυρία μου. Ευχαριστώ όλους σας ε, για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Ε, ξέρετε ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την ανταγωνιστικότητα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της. Όσον αφορά αυτά που ρώτησε ο κύριος Μπόνι ε, για τις προκλήσεις σε σχέση με το 5G. Έχουμε βέβαια και τους στόχους του 2025. Έχω, εκτός από τους τρεις στόχους που ανέφερα στην αρχή, έχουμε και τον στόχο ε, τη σύνδεση σε μένα, τουλάχιστον gigabyte, ε, σε όλους τους οικονομικούς ε, φορείς, την απρόσκοπτη ροή 5G, καθώς επίσης και το ποσοστό των 100 GB ανά δευτερόλεπτο. Είναι πολύ δύσκολο να, αυξηθούμε, να αυξήσουμε τα megabytes γιατί δεν έχουμε καλύψει καν τους στόχους για την ψηφιακή, για το ψηφιακό θεματολόγιο του 2020. Για το 5G θέλω να σας πω το εξή. Μερικές φορές ε, ή συχνά μάλλον μας ρωτάνε τι είναι καλύτερα το 5G, οπτικές ίνες, ε, ε, πού ακριβώς βρίσκεται το 5G. Βεβαίως το ελεγκτικό συνέδριο δεν είναι τόσο εξοικειωμένο με τα τεχνολογικά, αλλά εκείνο που γνωρίζουμε και που μπορούμε να πούμε είναι ότι το 5G δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τις οπτικές ίνες, να τις συμπληρώσει. Και οι οπτικές ίνες είναι η βασική υποδομή που είναι απαραίτητη για να μπορεί να λειτουργήσει και το σύστημα 5G. Εάν λοιπόν αυτό είναι απάντηση στην ερώτησή σας, εμείς αυτό μπορούμε να πούμε. Βεβαίως για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος του 5G ε, πρέπει να υπάρχει υποδομή και αργότερα βέβαια θα αναφερθώ ε, σε διάφορες λύσεις ε, τις οποίες επέλεξαν τα κράτη-μέλη. Γιατί θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την ευρυζωνικότητα. Ως εκ τούτου κάθε κράτος μέλος ε, έχει τη δική του την αρμοδιότητα να επιλέξει αυτό που επιθυμεί και με τα διάφορα παραδείγματα και θα αναφερθώ στην επόμενη ερώτηση για τις στρατηγικές μπορείτε να δείτε ότι το κάθε κράτος μέλος μπορεί να αναπτύξει τη δική του στρατηγική. Έχουμε το παράδειγμα των πέντε κρατών μελών που επισκεφτήκαμε. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία επέλεξαν να, έχουν, να υιοθετήσουν ένα μοντέλο όπου θα ε, επενδύσουν στο εφιστάμενο δίκτυο χαλκού. Ε, έχει πολύ καλές ε, γραμμές από χαλκό, οι παλιές τηλεφωνικές γραμμές που είναι βέβαια η πιο φτηνή τεχνολογία, όμως δεν επιτρέπουν υψηλότερε ταχύτητες. Άρα δηλαδή ακόμα και αν ε, χρησιμοποιηθεί αυτή η νέα τεχνολογία ε, και έτσι μπορείτε να αυξήσετε και με την παλιά δηλαδή ε, μπορείτε να ε, αυξήσετε μέχρι τα 100 MB δευτερόλεπτο αν είναι λίγοι οι χρήστες. Αυτό είναι το όριο όμως γιατί οι παλιές τεχνολογίες βασίζονται στον αριθμό των χρηστών όσο περισσότεροι χρήστες τόσο πιο πολύ μειώνει τη ταχύτητα. Έχουμε ένα παράδειγμα που ένα κράτος μέλος επιλέγει μια τεχνολογία ένα άλλο παράδειγμα είναι η Ιταλία, γιατί και εσείς αλλά και η κυρία Βιρκόνεν ε, ζήτησαν να αναφέρω ε, καλά παραδείγματα. Πρέπει να σας πω, ο στόχος της έκθεσης δεν είναι να αξιολογήσουμε εμείς τις επιδόσεις των κρατών μελών, αλλά έχουμε πέντε ε, κράτη-μέλη, είναι ενδεικτικά ως παράδειγμα και στο γράφημα θα δείτε ότι και 28 και 28 κράτη-μέλη έκαναν πρόοδο. Αν δείτε ποια ήταν η κατάσταση το 11 και ποια είναι το 17 θα διαπιστώσετε ότι όλοι προχώρησαν. Τώρα το ποιος ε, κατάφερε τη μεγαλύτερη βελτίωση Νομίζω στο γράφημα βλέπετε με απόλυτη σαφήνεια ότι η Ιταλία είναι ένα κράτος μέλος όπου η πρόοδος πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Αυτό το εντοπίσαμε και εμείς με τον έλεγχο. Και είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα απαντώντας στην ερώτησή σας. Και γιατί λόγω της επιλογής που έκαναν τα κράτη-μέλη ως προς τη στρατηγική τους, το πώς δηλαδή να αναπτύξουν το δίκτυο και κατά κάποιον τρόπο μπορείτε να συγκρίνετε την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, όπου υπήρχε σε όλες αυτές τις χώρες ε, ε, υποδομή με χαλκό, αλλά σε αντίθεση με τη Γερμανία, η Ιταλία επέλεξε ένα άλλο επενδυτικό μοντέλο. Ε, άρα δηλαδή επέλεξαν τελείως διαφορετικό επενδυτικό μοντέλο και αποφάσισαν να επενδύσουν πλήρως σε οπτικές σύνες. Με αυτήν λοιπόν, με αυτές τις ε, οπτικές ίνες έκαναν ένα, σαν ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την κάλυψη και κυρίως ε, στην ε, υποδομή η οποία ειλικρινά άλλαξε, άλλαξε ριζικά σε σχέση με αυτό που υπήρχε παλαιότερα. Κάτι άλλο που αφορά στην ερώτησή σας σχετικά με την ε, προσβασιμότητα για, τις, ε, για την Ήπεθρο και τις γεωργικές περιοχές. Πολύ σημαντικό αυτό το ερώτημα γιατί έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε και την ευρύτερη εικόνα η οποία έχει σχέση και με τις ε, πηγές χρηματοδότησης αυτής της πολιτικής ευρυζωνικής κάλυψης. Αυτό πρέπει να είναι και το σημείο κίνησης. Οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι όπως σας είπα ε, περίπου 250 δις εκτιμά η Κομισιόν ότι χρειάζεται για να επιτευχθεί ο στόχος. Αλλά από πού προέρχονται τα χρήματα. Προέρχονται κυρίως από ιδιώτες, ε, παρόχους και η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εθνική και η περιφερειακή είναι πάρα πολύ περισμένη Αν δείτε λιγάκι τα στοιχεία που αναφέρονται στην έκθεση, 15 δις, ε, τα μισά είναι ε, επιδοτήσει και τα άλλα δάνεια. Είναι περίπου το 6% του συνόλου. Και αυτό εξηγεί εν μέρη την ερώτησή σας το γιατί υπάρχει τόσο περιορισμένη προσβασιμότητα και τόσο περιορισμένη κάλυψη. Απλά και μόνο διότι ο ιδιωτικός τομέας ενδιαφέρεται για το κέρδος και όπου δεν υπάρχουν κερδοφόρες ε, περιοχές δεν επενδύει. Και εκεί βεβαίως ε, η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον γίνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Σε ορισμένε περιπτώσει που αναφέρονται στην έκθεση, υπάρχει μια περίπτωση ενό δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπου τα κονδύλια δεν χρησιμοποιήθηκαν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, γιατί δεν διοχετεύτηκαν στι ε, ε, περιοχέ που χρειαζόντουσαν πραγματικά αυτήν την ε, επένδυση. Όσον αφορά ε, θέματα ανταγωνιστικότητας και κανονιστικά ερωτήματα, αυτά ε, δεν σχετίζονται με το δεύτερο ερώτημα της κυρίας Βιρκούνεν, ότι θέλω να πω το δεύτερο σημαντικότερο θέμα μετά τη χρηματοδότηση. Ξέχασα να πω σε σχέση με τη χρηματοδότηση ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι τα κράτη-μέλη ε, έκαναν μια σωστή αξιολόγηση ε, των κονδυλίων που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτές τις ε, προκλήσεις. Τα περισσότερα κράτη-μέλη που επισκεφτήκαμε έκαναν αυτή την ανάλυση, κάποια άλλα πάλι όχι. Είναι λοιπόν απόλυτα σαφές ότι αν δεν έχεις κάνει μια σωστή ανάλυση για το πόσα κονδύλια χρειάζεσαι, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Κατόπιν, όσον αφορά το κανονιστικό και το ανταγωνιστικό πλαίσιο, αυτός ε, είναι ο δεύτερος, ίσως όχι και τόσο αμεληταίος παράγων, γιατί όταν υπάρχει ανταγωνισμός, αναμφίβολα, δημιουργούνται δυσκολίες για νέους παρόχους, ε, εφόσον αυτοί επιθυμούν ε, να δραστηριοποιηθούν. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στη Γερμανία, όπου ήταν δύσκολο για τους ε, καταναλωτές να φύγουν από έναν πάροχο, ε, ήταν δύσκολο να, για κάποιους νέους παρόχους να ε, στην αγορά. Στην Ιρλανδία υπήρχαν και κάποια θέματα ε, που έχουν σχέση με τον ανταγωνισμό. Εμείς όμως διαπιστώσαμε ότι το κανονιστικό και ανταγωνιστικό πλαίσιο ήταν αποδεκτό. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση οικονομικών χρηματοδοτικών εργαλείων, ένα που είναι πολύ ευπρόσδεκτο εργαλείο είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρυζωνικότητας. Το σημαντικότερο για μας και το ελεγκτικό συνέδριο είναι να υπάρχει αποτελεσματική αξιολόγηση χρήση των κονδυλίων. Και αυτό λαμβάνεται υπόψη και στις συστάσεις που καταθέτουμε. Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης ε, στην ε, υψηλή ταχύτητα στις ε, χώρες Μπενελούξ και μου έχει τεθεί το ερώτημα κατά πόσον υπάρχουν κράτη-μέλη όπου η ύπεθρος να είναι πιο εξελιγμένη, πιο ανεπτυγμένη από άλλες περιοχές. σχεδόν παντού εντοπίσαμε προβλήματα στην ύπεθρο, αλλά στις ε, χώρες Μπενελούξ και σε μικρές χώρες όπως η Μάλτα. Εκεί υπάρχουν πιο αναπτυγμένες ε, υπαίθριες περιοχές. Αυτό βέβαια εξηγείται και από το μέγεθος της χώρας. Σας είπα γιατί είναι μικρότερες χώρες και εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να αναπτυχθεί η υποδομή. Νομίζω ότι προς το παρόν ε, κάλυψα όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ αν ε, μπορούσαμε εμείς να οργανώσουμε ε, την χώρα μας, θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια τόσο μεγάλη πρόοδο όπως τον Benelux. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς επένδυσε η Ιταλία στις οπτικές ίνες στο Νότο. Είναι εξαιρετικό. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα υπάρχουν επαρκείς επενδύσεις σε οπτικές ίνες σε όλες τις χώρες μας. Και μάλιστα δεν μπορώ να φανταστώ τη Βόρεια Σουηδία, τη Βόρεια Φιλανδία που δεν ε, είναι και μεγάλος ε, ο πληθυσμός εκεί. Μπορώ να φανταστώ ότι στο Ελσίνκι ε, και στο Μάλμο, στην Κοπενχάγη θα υπάρχουν καλύψεις, αλλά σε αυτές τις αγροτικές περιοχές και ιδίως στη Γαλλία θα είναι πρόβλημα αυτό. Γιατί από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας των επενδύσεων για τις ιδιωτικέ εταιρείε αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τα πολύτιμα σχολιά σας και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο γιατί είχε έρθει και ο χρόνος ολοκληρώσαμε την έκθεση σχετικά με τι υποδομέ ευρυζωνική σύνδεση υψηλή ταχύτητα και πάμε στο Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτο 2019. Όλα τα τμήματα. Η συγητή είναι ο Γιάννη Γκάιερ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι εδώ εργάζομαι με μεγάλη χαρά. Βέβαια είμαι και αντιπρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών και κατόπιν τούτου υπάρχουν κάποια θέματα που δεν αφορούν, αφορούν άμεσα αυτή την Επιτροπή, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να τα εξετάσουμε. Όπω παραδείγματος χάρη ε, γνωμοδότηση για το γενικό προϋπολογισμό. Ε, θα ήταν ίσως ε, ωραίο και ενδιαφέρον να υπήρχαν άλλοι συνάδελφοι να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Ε, θα ήταν χρήσιμο να μοιραστούμε λιγάκι τις γνώσει μα και θα χαιρόμουν πάρα πολύ να μην είμαι αναγκασμένη σε αυτήν την επιτροπή να ασχολούμαι και με τον προπολογισμό. γιατί ξέρετε εγώ ήρθα στην Επιτροπή βιομηχανία, για να μην κάνω αυτά που κάνω έτσι καλώ σε άλλε επιτροπές τέλος πάντων, μπας περιπτώσει η γνωμοδότηση της Επιτροπής μας προς τον Γενικό Συγητή κατ' ουσίαν λαμβάνει την εξής μορφή ε, στέλνουμε μια επιστολή στον πρόεδρο. Αυτή την συστήσαμε από κοινού, κύριο Μπουζίκα και εγώ και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά και τους ε, σκιώδεις εισηγητές του πρόεδρου μας. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Βιομηχανίας στον προϋπολογισμό του 2019, η γνωμοδότηση αυτή ε, προσανατολίζεται σε όλα αυτά που γνωρίζετε από τα παλαιότερα έτη. Δηλαδή, καταρχήν, η διαδικασία του προπολογισμού γίνεται ως εξής. Το Μάιο η Επιτροπή καταθέτει ένα σχέδιο, αυτό πάει στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο αυτήν την πρόταση κατά κανόνα την περικόπτη και ριζικά. Ε, τα επιχείρηματα δεν είναι πάντα πιστικά, γιατί γίνεται αυτό. Και ένα από τα πράγματα που καλείται να κάνει κάθε εισηγητής του προϋπολογισμού ή συντάκτης κάποιας γνωμοδότησης είναι να επαναφέρει τα θέματα και τα ποσά σε αυτά που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς το κάναμε αυτό. Κάτι άλλο, το οποίο επίση γίνεται εδώ και πολλά χρόνια. Οι γραμμές του προϋπολογισμού που έχουν περικοπεί αφορούν ε, τις εγγυήσει ε, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο ε, Στρατηγικών Επενδύσεων. Οι περικοπές αυτές θα έπρεπε να επανέλθουν στο σημείο που ήταν πριν εμφανιστεί το ΕΦΣΥ. Ας δούμε λιγάκι το ιστορικό. Στην Επιτροπή αυτή σχεδόν κανείς δεν διαφωνεί με την χρησιμότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Σίγουρα η δική μου η πολιτική ομάδα δεν το πράττει αυτό. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το FC είναι μια δεξαμονή δάνειοδότησης. Η κυρία Ιβάνοβα αναφέρθηκε και εκείνη στη μελέτη της. Είναι ένα εργαλείο δανειοδότησης, αλλά για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος ε, ε, κόκκινων δανείων, έχουμε στον προϋπολογισμό μας ε, ποσά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν δεν μπορούν να αποπληρωθούν δάνεια. Αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι λυπηρό γιατί τα κονδύλια τα οποία είχαν προβλεφτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κονδύλια αυτά έχουν ληφθεί από προγράμματα τα οποία έπρεπε όμως να υπάρχουν. Πρόκειται λοιπόν για δύο γραμμές του πεπλογισμού που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα αυτήν την Επιτροπή. Είναι το κοινό ερευνητικό πρόγραμμα αφενός και κατά δεύτερον το εργαλείο Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να επαναφέρουμε ε, τα κονδύλια σε αυτές τις δύο γραμμές ε, στο ύψος που υπήρχαν. Και το τρίτο που θέλω να πω με την ιδιότητά μου ως μόνιμος εισηγητής για τους εξωτερικούς οργανισμούς στον Γενικό Προπολογισμό. Ε, γι' αυτό λοιπόν θελήσαμε να ρωτήσουμε τους εξωτερικούς οργανισμούς ε, κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μετά από αυτές τις ερωτήσεις προσθέσαμε ε, τα ποσά που επιθυμούν οι οργανισμοί αυτοί. Ενίσα, ΕΣΑ και άλλοι οργανισμοί. Αυξήσαμε τα κονδύλια για αυτούς τους οργανισμούς για να μπορούν και αυτοί οι οργανισμοί να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Σε γενικές γραμμές λοιπόν ο προϋπολογισμός από, την, από το πρίσμα αυτής της ε, Επιτροπής ε, καταλήγει στο ότι στο 1α αυξήθηκαν τα ποσά, στον, στο πρόγραμμα ορίζοντας επίσης ε, για την προστασία του κλίματος αυξάνονται τα κονδύλια κατά 20%. Αυτά όλα συμβάλλουν έτσι ώστε να επιδιωχθούν οι πολιτικοί στόχοι τους οποίους ε, επιθυμούμε. Το σχέδιο της γνωμοδότησης σας έχει διατεθεί και όταν θα έχετε δώσει τη συνένεσή σας, αυτή η γνωμοδότηση θα αποτελεί υλικό για τον γενικό εισηγητή, το συνάδελφό μου. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γκάια. Η Επιτροπή Ήτρε ε, προετοιμάζει γνωμοδότηση για την ε, Επιτροπή Προϋπολογισμού, η οποία είναι αρμόδια για το θέμα. Και ο αξιόλογος συνάδελφός μου, μάλλον η συνάδελφή μου, θα έχουν δύο λεπτά στη διάθεσή τους ως εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων για να εκφράσουν τις απόψεις τους ή για να υποβάλουν ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον εκπρόσωπο των ομάδων, ο κύριος Σαλίνη από το ΕΛΚ πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το σχεδιάγραμμα του ε, ε, εισηγητού Γκάγερ συμπίπτει με τις προτεραιότητες που διαπιστώνουμε κι εμείς. Οπωσδήποτε ένα από τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ευαισθησίας, μια και μιλάμε για την Επιτροπή βιομηχανία, αφορά την ε, συνέχεια που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα ε, στην προσοχή που δίνεται, η σωστή και ορθώς δίνεται αυτή η προσοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικό ε, αποτέλεσμα που διασφαλίζεται από το πρόγραμμα, αλλά την σχέση ε, ανάμεσα σε αυτά που πηγαίνουν ε, στο ε, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και αυτά τα οποία θα αφαιρεθούν από άλλα προγράμματα, τα οποία με τη σειρά τους όμως έχουν δείξει εξαιρετικά αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά ας πούμε τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe η Επιτροπή μας όπως και η Επιτροπή Τραν γιατί συζήτησα και με αυτήν την Επιτροπή Μεταφορών δηλαδή τα θέματα αυτά ε, και για μας το πιο σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ε, ε, προτάξουμε ως Επιτροπή Βιομηχανίας είναι ακριβώς η διασφάλιση ε, ότι θα υπάρξει ένα καλό εργαλείο υποστήριξης της καινοτομίας ε, που, και της βιομηχανίας που θα δείχνει ακριβώς ότι υπάρχει μια ισχυρή ρωμαλαία βιομηχανική πολιτική η οποία μπορεί να ε, προωθήσει την Ευρώπη. Ο προϋπολογισμός που προτείνεται είναι ικανοποιητικός και κατά τη δική μου άποψη, αλλά εάν θέλουμε πραγματικά να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, είναι να, να βεβαιωθούμε ότι μέσω αυτού του προϋπολογισμού οι βιομηχανικές πολιτικές θα πάρουν ακριβώς την κεντρική θέση που τους αρμόζει. Είναι σημαντικό να δούμε λοιπόν πώς θα διασφαλίζονται οι επενδύσεις και ε, αυτοί που ασχολούνται με την βιομηχανία να μην ε, έχουν διαρκώς νέες υποχρεώσεις. Αυτά όσον αφορά ε, τα θέματα αυτά λοιπόν συμφωνώ ότι η αναφορά στην ε, διαστημική πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, η αναφορά στο GSA της Πράγας επίσης ε, είναι σημαντική. Τα υπογράμμισα και εγώ αυτά στη δικιά μου γνωμοδότηση για την Επιτροπή Μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σαλίνη. Απ' την Άλντε, εξ ονόματος του κυρίου Ντομινίκ Ρικέ, Ευχαριστούμε πολύ τον ε, κύριο ε, τον εισηγητή, τον κύριο Γκάγερ. Όσον αφορά τώρα τα, ε, την, ε, τα προγράμματα. Ε, εμείς θεωρούμε ότι τα προγράμματα προστιθέμενης αξίας, αυτά δηλαδή που προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να προωθηθούν και τα λοιπά. Συμφωνούμε με την γνωμοδότηση. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Επόμενος... Ο κύριος Σιλικιώτης, ο έγκριτος Παρακαλώ κύριε Σιλικιώτη. ε, αρχικά θέλω να ευχαριστήσω τον Σεραφόν τον Γκάιερ ε, για τη συνεργασία που είχαμε για την πρόθεσή του να υποστηρίξει και τι σημαντικότερε θέσει όλων των πολιτικών ομάδων. Ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα που έχει η Επιτροπή μα είναι η συνδιαμόρφωση του πολιτισμού για τα κονδύλια που αφορούν θέματα των δικών μα αρμοδιοτήτων. Και εκεί θα επικεντρωθώ. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ω ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, Βόρεια Πράσινη Αριστερά, καταθέσαμε διάφορε τροπολογίε προτείνοντα να ανακατανεμηθούν τα κονδύλια με στόχο να εξυπηρετούν καλύτερα οι ανάγκε τη κοινωνία, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και τη βιομηχανία, ιδιαίτερα εκείνων των κρατών μελών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και είναι γνωστό ότι ιδιαίτερα στον Νότο υπάρχει μια διαδικασία αποβιομηχανοποίηση. Ιδιαίτερα όμω αρνητική κατά την άποψή μα είναι η πρόταση για επενδύσει στην άμυνα και την ασφάλεια, κάτι που σημαίνει περαιτέρω στρατιωτικοποίηση τη Ένωση. Και είναι γι' αυτό που με σχετική πρωτοβολία που έχουμε καταθέσει ζητάμε το κονδύλι που προορίζεται για δυναμική βιομηχανία να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παρόλο που οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι η ραχοκαλιά τη οικονομία ολόκληρη τη Ένωση, δυστυχώ τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν, ιδιαίτερα τώρα εν μέσω οικονομική κρίση, είναι πολλά και δυσβάσταχτα. Γι' αυτό είναι σημαντικό και αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τα κονδύλια για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διασφαλίζοντα ταυτόχρονα ποιοτικέ και αξιοπρεπεί θέσει εργασία. Ζητάμε λοιπόν την αύξηση των κονδυλίων που δίνονται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COSME, που στόχο έχει στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώ και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ορίζοντα 2020 για την έρευνα και την καινοτομία. Ζητάμε να αυξηθεί το ποσό που δίνεται για βελτίωση τη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, καθώ και το κονδύλι που δίνεται για γενικότερη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα με στόχο τη δημιουργία των νέων θέσεων εργασία με ενισχυμένα εργασιακά δικαιώματα. Εξίσου σημαντική είναι και η τροπολογία που έχουμε καταθέσει προτείνοντα να αυξηθεί το κονδύλι για την πρόθεση τη καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρησιών, καθώ και το κονδύλι που δίνεται για στήριξη τη έρευνα και ε, που οδηγά σε πύληση πολλών προβλημάτων τη κοινωνία. Τέλο, ε, να πω αγαπητοί συνάδελφοι ότι έχουμε καταθέσει μια τροπολογία η αύξηση του κονδυλίου που θα δοθεί για την πρωτοβουλία δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi for Europe, ώστε να καλυφθούν ανάγκε κυρίω των μικρών Δήμων και κοινοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιτευχθεί η γεωγραφική ισορροπία. Πρέπει να σα πω ότι επειδή ήμουν και ο διεισηγητή στο φάκελο για το Wi-Fi, ενώ έχει περάσει η θέση και είναι και εδώ ο συνάδελφο ο εισηγητή, ο συνάδελφο ο, ο, ο Κάρλο ε, Ζωρίνιο, ε, εν τούτης παρουσιάστηκε πρόβλημα στην έναρξη αυτού του προγράμματος γιατί αυτό το FES ΚΑΜ, ΦΕΡΣΕΒ οδήγησε χιλιάδες στα πέντε πρώτα δευτερόλεπτα από ό,τι ενημερώθηκαν να κάνουν αιτήσει. Εμεί ζητούμε να αυξήσει το κονδύλι και να μπορεί να υπάρξει στήριξη των μικρών Δήμων και των κοινοτήτων με μια γεωγραφική ισορροπία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Well, thank you very much. Uh, unfortunately... Σας ευχαριστώ. Δυστυχώς ε, υπερβήκατε το χρόνο επί δύο. Κύριος Ρούμπιχ, παρακαλώ, καταρχήν. Äh, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Αυτό που έχει σημασία είναι η στρατηγική την οποία ακολουθήσαμε κατά τελευταία χρόνια να ληφθεί υπόψη. Εγώ πιστεύω ότι η έρευνα και η ανάπτυξη για μας είναι απόλυτη προτεραιότητα και ως εκ τούτου θα ήταν σημαντικό να επιτύχουμε αποτέλεσμα από εκείνο το Συμβούλιο. Απευθύνομαι στον κύριο Σιλικιώτη. Ε, πολύ σωστά τα είπε. Ε, πράγματι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια και τέλος, όσον αφορά την Connecting Europe, το εργαλείο αυτό, ε, αποδείχθηκε ότι στο μέλλον πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Ε, για μένα αυτό πολύ σημαντική είναι η Silo and Vibe στρατηγική που έχει καταρτήσει η ΣΤΟΑ. Δηλαδή να υπάρχει καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς, να υπάρχει προστασία δεδομένων, να υπάρχει διαμεσολαβητής, να υπάρχει επιτροπή των περιφερειών. Νομίζω ότι οφείλουμε να καταρτήσουμε μια καλύτερη στρατηγική επικοινωνίας γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες εξοικονόμησης κονδυλίων αν υπήρχε εναρμόνιση όλων αυτών των οργανισμών, τουλάχιστον ως προς το διοικητικό σκέλος. Και πάρα πολλές ε, διατάξεις θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κατά πόσο μπορούμε να τις απλουστεύσουμε. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός του 2019 αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ως εκ τούτου οφείλουμε να ιεραρχήσουμε σωστά τα θέματα. Υπάρχουν μήπως ε, άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν σε αυτό το θέμα. Ωραία, έχω εγώ λοιπόν το λόγο. Θα ήθελα να τονίσω τη σημασία όλων αυτών των προγραμμάτων για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όπως υπόθηκε, η πλειονότητα αυτών των προγραμμάτων ε, είναι ε, τεχνικά πολύ ψηλά αναπτυγμένα και δεν ε, μιλάμε μόνο εδώ για τη χρηματοδότηση, αλλά πρέπει να πείσουμε και τις εθνικές κυβερνήσεις και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμπεριλάβουν τους εαυτούς τους αυτά τα προγράμματα, να συμμετέχουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα μεγάλα κράτη είναι αυτοί που δεσμεύονται περισσότερο σε όλα αυτά τα προγράμματα και το πώς ε, θα συμπεριλάβουμε και τα μικρά κράτη είναι απλό και λογικό. Θα πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα για όλες τις μικρές και μέσες επιχειρήσεις για συμμετοχή σε αυτά τα πολύπλοκα προγράμματα. Δηλαδή, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων, μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ μικρών και μεσανεπιχειρήσεων. επιχειρήσεων. Hope, Mr. Geyer. Ελπίζω λοιπόν, κύριε Γκάιερ, να πάρετε το λόγο και να βγάλετε ένα συμπέρασμα από τις παρατηρήσεις μας. Ελπίζω να κατανοήσετε μια πλήρη, να αντιληφθήκατε μια πλήρη εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ καλά τα γερμανικά σα ειλικρινά. Πολύ καλύτερα τουλάχιστον τα δικά μου τα τσέχικα και θέλω να σας πω ότι ε, δεν ε, είδα να διαφωνεί κανείς αλλά αν κάποιος θέλει κάτι να συμπληρώσει παρακαλώ τους συναδέλφους ε, να απευθυνθούν σε μένα. Εν πάση περιπτώσει ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία. Πολύ ωραία. Αυτά που είπατε ήταν πολύ ευσύνοπτα, θετικά και πολύ προοδευτικά καταδεικνύουν έτσι έναν δρόμο για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δηλώνουμε προθεσμίες. Έτσι λοιπόν, να έχετε κατά νου τις προθεσμίες για την κατάθεση τροπολογιών. Πρόκειται για την 5η Σεπτεμβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή Ήτρε, 24 Σεπτεμβρίου. Και ψηφοφορία στην Αρμόδια Επιτροπή, δηλαδή την Επιτροπή Προπολογισμών, 8 με 9 Οκτωβρίου. Φέτος. Ας ελπίσουμε ψηφοφορία στην Ολομέλεια προβλέπεται για τον Οκτώβριο. Είναι σαφείς λοιπόν οι προθεσμίες. Υπάρχουν σχόλια. Όχι. Επομένως, θα μπορούσαμε να κλείσουμε το σημείο αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκάιερ. Να πούμε στο επόμενο σημείο. Δέσπιση του διαστημικού προγράμματο τη Ευρωπαϊκή ε, Ένωση και του Οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το διαστημικό πρόγραμμα. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το διαστημικό πρόγραμμα είναι ένα από του πιο σημαντικού φακέλου και καλύπτει το Γαλιλαίο και το Κορπέρνικου, την ε, επιτήρηση και του του διάστημα και την πρωτοβουλία GovSatcom. Οι έδρες των προγραμμάτων αυτών βρίσκονται σε διάφορα μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, ακόμη και στην Πράγα έχουμε την έδρα του οργανισμού, στην ε, πρωτεύουσα τη Πατρίδα. μου. Είμαι πολύ περήφανο λοιπόν. Τώρα εδώ θα προβούμε στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων. χωρί έγγραφο, θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον κύριο Σαλίνη, τον εισηγητή, από το ΕΛΚ, να πάρει το λόγο και να ανοίξει τη συζήτηση. Θέλω να τονίσω από την αρχή ότι έχουμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας. Πρέπει να ολοκληρώσουμε στις 5 και 4. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι Είμαστε πολύ λίγοι εδώ, οπότε πολύ λιγότερο από 45 λεπτά θα χρειαστούμε για το θέμα αυτό, παρότι, όπως πολύ σωστά υπενθυμίσατε, αποτελεί κεντρικό θέμα και κεντρικό σημείο της συζήτησής μας και της στρατηγικής μας, να πω καλύτερα, της κοινή ευρωπαϊκής στρατηγικής. Επιτρέψτε μου να πω ότι... Ε, βλέποντας την εργασία αυτή πρέπει να αναγνωρίσω ότι έχουμε μπροστά μας ε, σε λίγο την τελευταία χρονιά της θητείας μας και παρότι τιμωρήθηκε, όχι απλώς επικρίθηκε η Ευρώπη ε, σε εκλογικές διαδικασίες πρόσφατα, παρόλα αυτά θεωρώ ότι τούτο εδώ είναι ένα από τα προγράμματα που δείχνουν τη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και το λέω έτσι με ε, πολιτική συνείδηση. Τα θέματα είναι πάρα πολλά. Ο χρόνος ε, για να προετοιμαστεί αυτό το πρώτο προσχέδιο που έπρεπε να ολοκληρωθεί μέχρι αύριο. Ήταν πολύ λίγος ο χρόνος, λέω. Επομένως, εγώ θα επικεντρώσω την προσοχή μου σε δύο θέματα κυρίως. προσπαθώντας τουλάχιστον σε τούτη τη φάση να σεβαστώ την πρόταση που μας έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία κρίνουμε θετικά. Κοιτάξτε, δεν είναι ε, τρομακτική, έτσι, ρηξικέλευθη, ας πούμε, κατάσταση ή όποια ε, επανάσταση, αλλά παρόλα αυτά ε, είναι ικανοποιητική και μας δίνει την δυνατότητα βαθμίας διαπραγμάτευσης και επομένως ε, να ξεκινήσουμε με στόχους επιτεύξιμους και όχι με οράματα τα οποία δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, να υλοποιηθούν. Ε, η διακυβέρνηση πρώτα απ' όλα, governance, πρόκειται για κεντρικό κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, τρία θέματα, συν ένα τέταρτο, ε, το οποίο είναι ε, επίπεδο, Το πρώτο βεβαίω στοιχείο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω κυρίως και της Κομισιόν, να παίξει σημαντικό ρόλο, γιατί πρόκειται εδώ για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι επομένως σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να ε, ηγηθεί των εργασιών που αφορούν ε, την διαστημική στρατηγική. Πρώτος συνομιλητής της Επιτροπής είναι ακριβώς η GSA που έχει έδρα την Πράγα που θα πρέπει, ε, ε, θα αλλάξει το όνομα, γίνεται πλέον Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για το Διαστημικό Πρόγραμμα ε, και τρίτον η, βεβαίως η ΕΖΑ, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Ε, όσον αφορά την ε, τωρινή GSA, πιστεύω ότι θα πρέπει να της δοθεί ένα νέο, αν όχι ενισχυμένο πλαίσιο. Κάποιες αρμοδιότητες από νομική άποψη έχουν εκχωρηθεί, ενώ άλλες ε, έχουν δοθεί, ε, άλλες αρμοδιότητες έχουν δοθεί σε αυτήν την ε, υπηρεσία προς αντιπροσώπευση. Ε, θα πρέπει να δούμε ποιες ε, είναι ε, οι κύριες αρχές, οι core, tasks και επίσης με ποιο τρόπο νομικά παρέχονται αυτές οι αρμοδιότητες σε αυτή την υπηρεσία η ε, πιστοποίηση της ασφάλειας, ε, η security accreditation που δίνει η Κομισιόν στην ε, GSA, εγώ προτείνω μεταξύ αυτών να δοθεί η ασφάλεια, η οποία δεν αναφέρεται καν στην πρόταση της Κομισιόν, που όμως εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ κεντρική σημασία θέματα, θέμα ε, στα πλαίσια της διαστημικής ε, ε, στρατηγικής. Επίσης υπάρχουν και άλλες λειτουργίες και άλλες αρχές οι οποίες είναι σημαντικές. Μην ξεχνάμε ότι το άρθρο 101 προβλέπει την αναθεώρηση σε κάποια χρονική στιγμή των επιδόσεων της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων ε, και ε, ενδεχομένως ε, προβλέπεται και κάποια δυνατότητα αναθεώρησης των αρμοδιοτήτων. Επίσης, η εγγύηση ότι θα παράσχεται τεχνητή αλλά όχι μόνο υποστήριξη από την ε, Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία γιατί μίλης ότι έχει πολλές και ιστορικές ε, αρμοδιότητες αυτή η ε, υπηρεσία πριν ακόμα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν τέτοια να ενδυθεί των διαστημικών. Και έχουμε και ένα τέταρτο ε, πολυμερές ας πούμε εργαλείο που είναι τα, τα, τα κράτη-μέλη τα οποία θα μπορούσαν να αναλάβουν συγκεκριμένα θέματα, tasks από την Κομισιόν, στα πλαίσια δηλαδή μιας νέας συμπροταγωνιστικ... ενός νέου συγγνώμη, συμπροταγωνιστικού ε, ρόλου. Ε, και ε, για λόγους προετοιμασίας ε, των επόμενων σταδίων. Ο προϋπολογισμός τώρα. Ο προϋπολογισμός είναι σημαντικός, 16 δις ευρώ έχουν ταυτοποιηθεί ως συνολικός προϋπολογισμός για την διαστημική πολιτική, μοιραζόμενο δε μέσω Γαλιλαίου, Κοπέρνικου και του SATCOM και του ESSA για τον ε, Γαλιλαίο πάνω από 9,5 δις και συγγνώμη, 4,5 για τον, ε, ε, για τον Κοπέρνικο ε, ενώ για, το, ε, για τα επόμενα δύο προγράμματα GovSat το SSA ε, 50 εκατομμύρια ευρώ για τον καθένα νομίζω ότι είναι ανεπαρκές ε, το ποσό αυτό. Και πιστεύω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να διπλασιαστεί. Στο σύνολο υπάρχουν πολλά σημεία, 5-6 θεμελιώδους σημασίας. Λέω ότι η απόψη μεθοδολογική και ακριβώς λόγω της έλλειψης χρόνου για το πρώτο αυτό σχέδιο, γι' αυτό θεώρησα ότι δεν θα έπρεπε ακόμα και για το προσχέδιο να ξεκινήσω από τις προτεραιότητες αλλά να ξεκινήσουμε με βαθμιαία προσέγγιση έτσι ώστε σιγά σιγά να ε, συζητήσουμε τα ε, θέματα. Ε, όμως θεωρώ ότι στην αρχή ε, θα πρέπει ε, να ξεκινήσουμε με βάση αυτές τις έξι πρώτες μεγάλες προτεραιότητες, αυτές τις οποίες ανέφερα στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας, για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θέλω να ζητήσω από τους συναδέλφους Σκιώδης να σεβαστούν το χρόνο αγόρευσης των δύο λεπτών. Καταρχήν, Σα Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Αξιότιμα κύριε Σίγητα, χαιρετίζω την ε, ε, πρόταση να υπάρχει ένα νέο κανονισμός για το διάστημα. Εν τω μεταξύ τα διαστημικά προγράμματα έχουν γίνει αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής πολιτικής, θα εξελιχθούν περισσότερο στο μέλλον. Και είναι σημαντικό ε, σε έναν και μόνο κανονισμό ε, να έχουμε ε, την απαραίτητη νομοθεσία. Βεβαίως υπάρχει μια στρατηγική από πέρυσι και αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Μεταξύ άλλων έχουμε ένα μεγαλύτερο προπολογισμό για το διάστημα σε σχέση με το μέχρι τώρα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το έτοιμο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ικανοποίησε με τα 16 δις. Φαίνεται όμω ότι δεν είναι σίγουρο κατά πόσον τα κονδύλια αυτά θα χρησιμοποιηθούν ή αρκούν για την επίτευξη όλων των στόχων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμφωνώ απόλυτα με τον εισηγητή. Για μα, όπω και για τον ε, εισηγητή, είναι απόλυτη προτεραιότητα να διατηρηθούν τα προγράμματα Κοπέρνικος και Γαλιλαίο, ε, τα οποία αποφέρουν προ τη θέμενη αξία και είναι αυτά τα οποία κατέστησαν την Ευρώπη ανεξάρτητο παίκτη ανά τον κόσμο. Και τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν έτσι ώστε να ενισχυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρος ε, καινοτομιών. Κατά τα άλλα, το πρόγραμμα για το διάστημα θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω. Σε τελική ανάλυση ε, υπάρχουν και το θέμα των ε, υπολοιμάτων από το διάστημα. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και ως εκ τούτου ε, τα 250 εκατομμύρια δεν φτάνουν αυτά που έχουν προταθεί. Ο προπολογισμό ε, για το διάστημα ε, συνδέεται άμεσα με το Rising Europe. Το διάστημα χρειάζεται πάρα πολλές έρευνες, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν κονδύλια της τάξης των δις. Αυτό που βλέπω με κριτικό πνεύμα είναι είναι η πρόταση της Επιτροπής η ασφάλεια και η άμυνα να καταστούν καθοριστικό σημείο στην ε, περαιτέρω ανάπτυξη του διαστήματος. Ακόμα και αν είναι απαραίτητο και αυτονόητο να βελτιωθεί η υποδομή για να μην υπάρχουν πλέον κρίσεις, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα προγράμματα του διαστήματος είναι αστικής φύσης και ως τέτοια θα πρέπει να παραμείνουν. Ως εκ τούτου, για την μελλοντική διαμόρφωση των προγραμμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, θέματα κλιματικής αλλαγής, ε, συνδεσιμότητα, να ληφθούν υπόψη και στον προπολογισμό. Ένα άλλο βασικό στοιχείο του κανονισμού είναι η διαχείριση. Στην διαστημική πολιτική υπάρχει στενή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Διαστήματος όπως και με τον οργανισμό GNSS. Εμείς στην έκθεσή μας για το διάστημα αναφέρουμε ότι θα πρέπει οι αρμοδιότητες όλων αυτών των φορέων να είναι σαφέστερος από ό,τι μέχρι τώρα. Και όσον αφορά την ε, εμπορία των προγραμμάτων, την θέση εμπορία των προγραμμάτων Κοπέρνικος, η πρόταση Κομισιόν είναι ασαφής. Όμως θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια αν θέλουμε να ικανοποιήσουμε όλες αυτές τις προσδοκίες που υπάρχουν για προστιθέμενη αξία. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μπορώ να συνεργαστώ με τον εισηγητή και τον σκιώδη εισηγητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Πρόεδρος. Ε, ξεπεράσατε το χρόνο σας ή τον εξαντλήσατε, εν πάση περιπτώσει, αλλά όλα αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Κυρία Άννα Χταγκαλίων, επόμενη. Ναι, ευχαριστώ. ορίζω την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα. Νομίζω ότι εδώ θα συγχωνεύσουμε τις παλιές με τις νέες πρωτοβουλίες για το διάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει σημαντικό δυναμικό από το πρόγραμμα για να τονώσει την κοινοτομία, την ασφάλεια αλλά και τις οικονομικές δραστηριότητες ε, στους τομείς κατά αντί και μας βοηθά να ψηφοποιήσουμε περαιτέρω την οικονομία μας. Επίσης θα πρέπει να βελτιώσει και την παρακολούθηση των των ικανότητα παρακολούθηση κλιματική αλλαγή είναι ένα στοιχείο τη πρόταση που καλωσορίζουμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη και για την επίλυση των παγκόσμιων προκλήσεων. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν εκφράσει ε, σκεπτικισμό απέναντι σε κάποιες πτυχές της πρότασης, αλλά ε, σε ό,τι μεταφορά η πρωτοβουλία της Κομισιόν δίνει μεγαλύτερες ευκαιρίες ε, για να υπάρχει εξορθολογισμός και να δημιουργηθούν συνέργειες. Τους επόμενους μήνες θα έχω πολλές συνεδριάσεις και με ενδιαφερόμενα μέρη και εκπροσώπους του τομέα. Επομένως, περιμένω να υπάρχει περαιτέρω συνεργασία με τους κοιόδης αλλά και με τον εισηγητή για το φάκελο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις παρατηρήσεις σας. Ο κύριος ε, Κόχλητσικ είναι ο επόμενος, εγώ δηλαδή. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη σημασία όλων των προγραμμάτων που έχουν ε, απαριθμηθεί και συμπεριλαμβάνονται σε όλο το χώρο της ε, τεχνικής ανάπτυξης ε, είναι σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε να θεωρούμε ότι έχει ηγετικό ρόλο σε θέματα που αφορούν ε, και τα περιβαλλοντικά. Έτσι λοιπόν το Κοπέρνικους είναι πολύ εργαλείο όχι μόνο για τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και για τα όμορα κράτη. Υπάρχουν πολλά κράτη που θα ήθελαν να συμμετέχουν στο Γαλιλαίο. Mm. Αναπτύσσεται γρήγορα η υπηρεσία για, υπηρεσίες για το Γαλιλαίο. Έχουμε μέχρι τώρα 30 δορυφόρους. Επομένως αυτό θα πρέπει να ληφθεί όντως υπόψη. Τονίσατε κάποιος από εσά, η κυρία Κρέλ ιδίως, τόνισε κάτι που θέλω να πω και εγώ. Ότι πρέπει να σκεφτούμε και τη μη στρατιωτική χρήση όλων αυτών των προγραμμάτων. Η στρατιωτική χρήση είναι ένα τμήμα των συμφερόντων μας Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι θα πρέπει να διατηρούμε τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιούμε καταλήλως. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτά τα μεγάλα project δεν είναι τόσο εύκολο να συμμετέχουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ακόμη και στην τελευταία έκθεση της κυρίας Κρέλ, τονίσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτές οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, να συμμετέχουν σε όλα τα προγράμματα. Πιστεύω ότι είναι πολιτική απόφαση για το ποιο ε, θα αναλάβει πια καθήκοντα. Και θα πρέπει να δηλωθεί αυτό εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι τεχνικού χαρακτήρα αρμοδιότητες θα πρέπει να αναλαμβάνονται σε επίπεδο οργανισμών και δεν θα πρέπει να ενοχλούμε ε, αυτές τις ε, υπηρεσίες, αυτού του οργανισμού με εμπορικά ζητήματα. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει διαχωρισμό εμπορικών και τεχνικών καθηκόντων. Και φυσικά δεν μπορούμε να ε, υπερβάλλουμε, να αξιολογήσουμε μάλλον το τεράστιο αντίκτυπο και το τεράστιο δυναμικό αυτών των δραστηριοτήτων στο μέλλον. Αυτέ είναι οι παρατηρήσει μου ως εκπρόσωπο της ομάδας ΓΚΟΕ. Τώρα, ο δεύτερος γύρος για τα υπόλοιπα μέλη. Έχετε στη διάθεσή σας ένα λεπτό. Ο κύριος Μπλακολόπας καταρχήν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν ε, λίγους μήνες ε, ψήφισαμε στο Κοινοβούλιο το ψήφισμα για μια στρατηγική διαστημική για την Ευρώπη. Μεταξύ άλλων ζητούσαμε ένα προπολογισμό για το διαστημικό τομέα μεγαλύτερο από το σημερινό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις του τομέα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν έχει λάβει υπόψη το αίτημα αυτό από τα 12 δισεκατομμύρια πέρασε στα 16 δισεκατομμύρια ε, που προβλέπονται στο νέο πρόγραμμα. Επίσης, είχαμε ζητήσει να μεγιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των διάφορων διαστημικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που τώρα έχουμε μπροστά μας είναι μία πρόταση που συγχωνεύει τέσσερα από αυτά τα προγράμματα και φυσικά θα συμβάλλει σε αυτό το στόχο. Και ελπίζουμε όλα αυτά να συμβάλλουν στο να προωθήσουν την παγκοσμιακή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωση στον τομέα, να δημιουργήσουν μία πιο ισχυρή και καινοτόμο βιομηχανία και να εγγυθούν μία ασφαλή πρόσβαση ε, και ανεξάρτητη της Ένωσης στις επικοινωνίες μέσω δορυφόρου. Και Πιστεύω ότι και οι συνάδελφο Κωνσταντίνα και οι υπόλοιποι θα κάνουν τα κατάλληλα σχόλια και συνεισφορά για να πετύχουμε του στόχου αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει άλλος κανείς που θα ήθελε να καταθέσει εδώ τις ιδέες του. Σε αυτόν τον πρώτο εισαγωγικό γύρο. Όχι. Τότε να δώσουμε Καταρχήν το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον εκπρόσωπο από τη ΓΑΜΑ Ανάπτυξη. Συγγνώμη, δεν μπορώ να σας απαντήσω τσέχικα. Θα προσπαθήσω για την επόμενη φορά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας και την ευρία υποστήριξη που άκουσα σε την αίθουσα για την, ε, άποψη για την πρόταση της Κομισιόν. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια που πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Καταρχήν, όπως είπε ο εισηγητής, ε, δεν ε, παρουσιάσαμε κάτι επαναστατικό, απλώς μία εξέλιξη. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο, γιατί δεν θέλαμε να αλλάξουμε τα πάντα. Μην φτιάχνεις κάτι που δεν έχει χαλάσει. Αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή και πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί όπω είπε και ο κύριος Σελήνη, αυτό που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα είναι μια τεράστια επιτυχία και ε, θα πρέπει να είμαστε περήφανοι που μπορούμε να απτύξουμε αυτά τα προγράμματα. Το δεύτερο στοιχείο. Εξακολουθούμε να είμαστε φιλόδοξοι. Γιατί, όπως ε, μας είπατε, είμαστε φιλόδοξοι σε σχέση με το ποσό που θέλουμε να διαθέσουμε για το διαστημικό πρόγραμμα. Άκουσα τι είπε ο εισηγητής για το γνώσο ότι πρέπει να έχουμε περισσότερα χρήματα, ίσως για αυτά τα προγράμματα. Δεν διαφωνούμε βεβαίως, αλλά ε, ξέρετε, τώρα εσείς έχετε τον μπαλάκι στο γήπεδό σας να δείτε αν μπορείτε να κάνετε κάτι για το SSA και για το govsat.com. Όμω, ε, για το Κοπέρνικου και για τον Κελαιό αυτό που προβλέπετε είναι το ελάχιστο. Είναι λοιπόν δύσκολο να αφαιρέσουμε τα χρήματα από το Γαλιλαίους και το Κοπέρνικου ε, και να τα βάλουμε στον Govsat.com και στο SSA, στην ακριβή γνώση κατάσταση στο διάστημα. Βέβαια, δεν ξέρω από πού θα πρέπει να έρθουν τα χρήματα για αυτά τα δύο, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να αφαιρεθούν από τα Κοπέρνικου και Γκαλιλαίο. Έτσι λοιπόν, κάτι που πιστεύω είναι πολύ σημαντικό, είναι το θέμα τη διακυβέρνηση. Το είπατε κι εσεί. Είναι πάντοτε πολύπλοκο το θέμα, γιατί έχουμε εδώ ε, πολλού παίκτε, αλλά στο θέμα τη διακυβέρνηση θα έλεγα καταρχήν η Κομισιόν, βεβαίω, θα πρέπει να παραμείνει σημαντικό παίκτη. Και εμεί φυσικά θα πρέπει να σα εξηγούμε τι γίνεται με τα χρήματα του φορολογούμενου. Έτσι λοιπόν ε, είναι σημαντικό η Κομισιόν να έχει αυτό το ρόλο. Όμως ε, έχουμε εξαιρετική συνεργασία με την GSA και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και θα πρέπει να συνεχίσουμε. Θα πρέπει να εξορθολογήσουμε τη σχέση έτσι ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα ποιος κάνει τι και σε ποιες περιστάσεις. Και όπως αναφέρθηκε και από τον εισηγητή, είναι σαφές ότι η GSA θα παίξει ένα μεγαλύτερο ρόλο για την ασφάλεια, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τη διάσταση της ασφάλειας σε ένα διαστημικό πρόγραμμα και το θέμα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Έτσι λοιπόν η ασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη και να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό και στο μέλλον. Τέταρτο στοιχείο, στο οποίο θέλω να επιμείνω, είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ένα πολιτικό πρόγραμμα και θα παραμείνει πολιτικό πρόγραμμα, μη στρατιωτικό. Δεν μπορούμε όμω να γνωρίσουμε ότι υπάρχει και κάποια στρατιωτική χρήση, τουλάχιστον του Γαλιλαίου. Και ακούσατε και τη συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την πρόσβαση του Ηνωμένου Βασιλείου στο μέλλον στο Γαλιλαίο. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε εντελώ τη διαστασία αυτή, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σα με τα όσα είπατε ότι αυτό θα πρέπει να παραμείνει για μη στρατιωτική χρήση. Και πριν να να μακρηγορήσω ιδιαίτερα για τις μικρές και μισές επιχειρήσεις πρέπει να κάνουμε κάτι, είναι σημαντικό γιατί δεν μπορούμε ε, αυτά τα προγράμματα να τα φτιάχνουμε μόνο για τις μεγάλες εταιρείε. Ε, υπάρχει λοιπόν και ένα άρθρο που αναφέρεται στις μικρές και μισές επιχειρήσεις και τι πρέπει να κάνουμε στο διαστημικό τομέα και αν έχετε ιδέες για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το θέμα αυτό βεβαίως ευχαρίστως να ακούσουμε τις δράσεις αυτές. Και Παραμένω να δω και τις εξυπροτεραιότητες να ορίζονται από τον κύριο Σελήνη. Ξέρουμε τι δύο μέχρι τώρα. Αλλά σίγουρα θα θέλουμε να δούμε και τι υπόλοιπε με μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τα όσα πολύ θετικά μας είπατε. Νομίζω ότι είναι βιώσιμο στα προγράμματά μας, στο πρόγραμμά μας ε, να αναφέρουμε ότι και αυτοί που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ε, δεσμευτούν. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το, γύρω μας. Ωραία. Τώρα ήρθε η ώρα να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Σαλίνη, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Παρακαλώ κύριε Σαλίνη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτήν την πρώτη προσέγγιση και την πρώτη συζήτηση που είχαμε. Ε, να κάνω κάποιες ε, πρόσθετες αναφορές. Όπως αναφέρθηκε, ε, μια άλλη μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί κατά κάποιο τρόπο το βιομηχανικό, τη βιομηχανική, η βιομηχανική βαρύτητα που παρουσιάζει το πρόγραμμα αυτό, είναι η ε, η δραστηριότητα που σχετίζεται με το downstream. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ ασθενείς ε, όσον αφορά τους χρήστες αυτών των τεχνολογιών που αναπτύσσουν ε, εργαλεία ή applications, εφαρμογές όπως τα και smartphones κλπ και που προέρχονται από κυρίως μη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει ε, να αντιμετωπίσει αυτό αυτή την πρόκληση ενός ισχύρου upstream που ε, δίνει η διαστημική πολιτική έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ε, μια ε, ολοκληρωμένη βιομηχανική παραγωγή η οποία δεν θα υποστηρίζει μονάχα αλλά ε, θα έχει και μια ευρεία βιομηχανική βάση που θα χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες. Το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περηφάνεια κατά κάποιο τρόπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει βεβαίως να πραγματοποιηθεί και σε άλλα στοιχεία της στρατηγικής. Ας πούμε, access to space ε, δορυφόροι ε, που δεν ανέφερα προηγουμένως είναι ένα άλλο από τα στοιχεία προτεραιότητας από τον οποίο θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι και όσον αφορά το σημείο αυτό που είναι κεντρικό ε, στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Πολιτική έχουμε και εδώ πάρα πολύ μεγάλες ε, δυνατότητες και γνώσεις. Ε, θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε και το απαραίτητο νομικό πλαίσιο έτσι ώστε προτεραιότητα να δοθεί στους ευρωπαϊκούς δορυφόρους γιατί το σύστημα θα πρέπει να διατηρηθεί και από αυτή την άποψη. Θεωρώ ότι και από πολιτική απόψεω, εκτός από τη βιομηχανική απόψεω, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος, σωστή παρατήρηση με τον Govsat.com. Ε, ναι, θέλουμε να, να, το, ε, να το ενισχύσουμε, αλλά όχι ε, προζημίαν του Γαλιλαίου και του Κοπέρνικου γιατί η πρόκληση είναι μεγάλη και έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να δώσουμε δυνατότητες στον, στα δύο προγράμματα αυτά, Κοπέρνικο και Γαλιλαίο, έτσι ώστε, ε, μεταξύ άλλων βέβαια, έτσι ώστε να αναπτύξουμε νέες ε, δραστηριότητες ε, και να δώσουμε χώρο αυτή, σε αυτή τη διαστημική πολιτική. Give space to a space. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πρώτο γύρο συζητήσεων για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα λοιπόν να ε, ολοκληρώσω λέγοντας ότι ε, μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, 6 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι τροπολογίες. Η μελέτη των τροπολογιών θα γίνει την 9η Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία στην Ήτρε την 5η Νοεμβρίου. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια ε, δεν είναι ακόμα ε, γνωστή. Θα δούμε είτε το Δεκέμβρη είτε ε, τον Ιανουάριο. Αυτά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορούσε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα από αυτά που απασχολούν την Επιτροπή μας. Ωραία, τελειώνουμε λοιπόν με την εξέταση του σημείου 6 και περνάμε, περνάμε στο επόμενο σημείο. Δηλαδή, Σχέδιο σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου για τη σύνευση εξ ονόματο τη Ένωση τη Συμφωνία Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και του Βασιλείου του Μαρόκου για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη συμμετοχή του Βασιλείου του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς έρευνας και καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου, το επωνομαζόμενο πρίμα. Ίσως να πω ε, εξ αρχής ότι το βασίλειο του Μαρόκου στη δεκαετία του 70 ε, ζήτησε να έχει πρόσβαση σε αυτές τις διαδικασίες. Τότε είχε, ε, δεν είχε γίνει δεκτή, γιατί δεν ήταν ευρωπαϊκή χώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι ανοιχτή στις ευρωπαϊκές χώρες. Και μόνο. Ωστόσο, το Μαρόκο, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάντοτε με το Μαρόκο στενές σχέσεις. Και ξέρετε ότι είναι και πολύ ε, οι Ευρωπαίοι και οι Βέλγοι μαροκινής καταγωγής που ζουν στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες συγκεκριμένα. Το πρίμα ε, είναι εταιρική σχέση ε, μεταξύ δημοσίων φορέων και αφορούν ε, κυρίως και αφορά κυρίως την ασφάλεια όσον αφορά το νερό και τα τρόφιμα στην περιοχή της Μεσογείου. Και επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά, είναι σημαντική και η συνεργασία. Ε, το ε, πρόγραμμα Πρίμα ε, βλέπει τη συμμετοχή πολλών μεσογειακών γειτονικών χωρών και για να γίνει δυνατή η συνεργασία έπρεπε να υπογραφούν μια σειρά επιστημών και τεχνολογικών συμφωνιών συνεργασίας με τις συμμετέχουσες τρίτες χώρες μεταξύ των οποίων και το Μαρόκο. Ε, εδώ λοιπόν έχουμε τη συμφωνία με το Μαρόκο έτσι όπως ε, προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και που αφορά ένα διευρυμένο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας όσον αφορά το νερό και τα τρόφιμα. Θα ήθελα να σας πω ότι τα επόμενα 15 λεπτά θα τα αφιερώσουμε στην συζήτηση αυτή και ο κύριος Σαλίνη ε, θα αντικαταστήσει τον εισηγητή κύριο Άλτο Πατριτσέλο. Θέλετε να πάρετε το λόγο λοιπόν κύριε Σαλίνη. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ τον συναδελφό Πατριτσέλο. Έτσι λοιπόν θα διαβάσω το σημείωμα του εισηγητή. Ζητώ συγγνώμη από την Προεδρία, αλλά αμέσω μετά θα πρέπει να εγκαταλείψω την αίθουσα. Έτσι λοιπόν απλώς ε, θα διαβάσω την έκθεση που προτείνει ο συνάδελφος η εταιρική σχέση για την έρευνα και τη δημοκρατία στην περιοχή της Μεσογείου Πρίμα είναι η πρώτη δημόσια σύμπραξη μεταξύ φορέων του δημοσίου ε, και ε, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα βάσει το άρθρο 185 και ε, θέλει να ομαδοποιήσει τις ικανότητες έρευνας ε, της Ένωσης και των χωρών της Μεσογείου που συμμετέχουν προκειμένου να υπάρξει ανάπτυξη και νέες λύσεις που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια, την βιωσιμότητα των συστημάτων προμήθειας και διαχείρισης του νερού και αγροδιτροφικών προϊόντων. Στόχος είναι να συντονίσει και να ενισχύσει τα εθνικά προγράμματα έρευνας και κοινοτομία στους τομείς αυτούς, ε, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και αποτελώντας ε, ε, παράδειγμα επιστημονικής διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πλαίσιο που θέτει τη Μεσόγειο ε, στην πρώτη σελίδα λόγω των μεταναστευτικών φαινομένων. Ε, θέλουμε καταρχήν να έχουμε μια βέλτιστη πρακτική για να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε της μετανάστευσης και όχι μόνο για να καταπολεμήσουμε τα αποτελέσματα καθιστώντας την περιοχή της Μεσογείου πιο αηφόρο και σταθερή. Στη σημερινή κατάσταση 19 χώρες ε, ε, από κοινού ε, συμμετέχουν, 11 είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 3 χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα 2020 και 5 τρίτες χώρες με τις οποίες η Ένωση πρέπει να συνάψει διεθνείς συμφωνίες επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 της απόφασης. Η συμφωνία με το Μαρόκο ε, ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευση σε αυτό το πλαίσιο. Δεν θα μπω ε, σε θέματα που αφορούν ε, τώρα τη διένεξη του Μαρόκου με τη Δυτική Σαχάρα, θεωρώντα ότι αυτό το θέμα, αν και αποτελεί πολύ σημαντικό θέμα για γεωπολιτικό για την περιοχή, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο τη δική μα κοινοβουλευτική επιτροπή. Έτσι λοιπόν ε, ε, δέχομαι, υποδέχομαι θετικά την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας συνιστώ να εγκρίνετε τη συμφωνία. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 11η Ιουλίου και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα 3η Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία και ιδίως τον Αντρέ για την συνεχή υποστήριξη. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα ακολουθήσουν τώρα οι σκιώδεις συγητές. Ο πρώτος, ο οποίος είναι παρόν, η κυρία Τόγια. Παρακαλώ, κυρία Τόγια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την τελευταία διαβεβαίωση σχετικά με την πρωτοβουλία που πρόκειται να ληφθεί και το λεφτό έχοντας ε, παρακολουθήσει όλη αυτή την εξέλιξη και τη διαδικασία τις δυσκολίες ε, που υπήρχαν στη Μεσόγειο. Ε, οι πρωτοβουλίες ε, ήταν συγκαλυμμένες και νομίζω χάρη της παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όχι μόνο της δικής μου παρέμβασης, αλλά γενικότερα του Κοινοβουλίου, προάγαμε μια συζήτηση στο Στρασβούργο, ζητήσαμε από τον Επίτροπο να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Είναι λοιπόν μια από τις περιπτώσεις εκείνες όπου πραγματικά το Κοινοβούλιο έδειξε με ποιήση ότι μπορεί να αναλάβει οι πρωτοβουλίες και δείξαμε ότι είναι είναι σημαντικό να υπάρχει σχέση και με άλλες χώρες και ότι ο καθένας ε, να προσφέρει κάτι, να υπάρχει μια ε, πρωτοβουλία και για χώρες οι οποίες ε, δεν είναι ιδιαίτερα πρικισμένες, δεν έχουν πάρα πολλούς πόρους. Όπως είπε λοιπόν και ο εκτελών χρέη του εισηγητή, το θέμα δεν είναι μόνο ότι πράγματι είναι πολύ σημαντικό το θέμα των υδάτων του περιβάλλοντος, ε, οι επιπτώσεις που υπάρχουν από όλα αυτά στην ειρήνη και στην ανάπτυξη. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή η δουλειά είναι ουσιαστική και οι ευρωπαϊκές χώρες ε, ε, οι οποίες έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία βλέπουν ότι ακολουθούν και άλλες που τις στηρίζουν. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή πρωτοβουλία και νομίζω ότι πρέπει να τη στηρίξουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα αυτό. Εκπρόσωπος της Κομισιόν. Αντρέα Καρενιάνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρο, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας και στα μέλη αυτής της Επιτροπής για την υποστήριξη που προσέφεραν σε αυτή την πρωτοβουλία και θα ήθελα να επαναλάβω τα βασικά χαρακτηριστικά γιατί δεν είναι απαραίτητο να μπούμε σε λεπτομέρειες. Ο εισηγητής εξηγεί ότι πρόκειται για μια περιφερειακή μεσογειακή πρωτοβουλία. Είναι η πρώτη του είδους που αφορά σε εταιρική σχέση ανάμεσα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες που έχουν ήδη προσχωρήσει στον ορίζοντα 2020 και τρίτες χώρες με ακτές στη Μεσόγειο. Το τρίτο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω είναι η σημασία αυτής της πρωτοβουλίας. Ε, στόχος είναι να προκύψουν καινοτόμε λύσεις. Δεν πρόκειται τόσο για τη συνεργασία ανάμεσα σε χώρες, αλλά για τη συνεργασία επιστημονικών κοινοτήτων να ε, συνταχθούν ε, πόροι ερευνητές για ένα, μια βασική πλουτοπαραγωγική υπογή που είναι τα τρόφιμα και ε, το νερό και τα γεωργικά τρόφιμα. Διαχείριση λοιπόν όλων αυτών των πόρων και των συστημάτων. Η πρωτοβουλία ξεπερνάει το θέμα των υδάτων και των ε, γεωργικών τροφίμων γιατί αντιμετωπίζει και άλλες προκλήσεις όπως την κλιματική αλλαγή. Πώς μπορούν να αμβληθούν οι επιπτώσεις ε, από την κλιματική αλλαγή. Αντιμετωπίζονται επίσης και άλλες προκλήσεις όπως είναι η μετανάστευση και βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι κοντά στις ανάγκες των πολιτών. Δηλαδή ε, προκύπτουν ή ζητούνται συγκεκριμένα επιστημονικά αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα συνεργασίας επιστήμης και διπλωματίας. Συνεργαζόμαστε επίσης όρις με τους ε, διεθνείς εταίρους μας. Το Μαρόκο είναι ένας από αυτούς τους εταίρους. Το Μαρόκο έχει συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση αυτών των πρωτοβουλειών από τότε που συνελήφθησαν το 2012 και το Μαρόκο είναι πρόθυμο να συνεισφέρει και οικονομικά στην υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλειών και ακολουθεί μετά από άλλες χώρες ε, αφρικανικές και χώρες της Μέσης Ανατολής χώρες όπως η Αλγερία, ο Λίβανος, η Ορδανία και η Αίγυπτο χώρες οι οποίες έχουν ήδη διαπραγματευτεί και έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Στην περίπτωση του Μαρόκου χρειαζόμαστε ακόμα τη συνένεση, συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, αλλά είμαστε ε, αισιόδοξοι ότι ε, τα λάβουν όλοι υπόψη τους τα ωφέλη που μπορούν να προκύψουν για τους πολίτες αυτών των κρατών. Ε, τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω κάποιες παρατηρήσεις μου. Το πρόγραμμα Πρίμα ξεκίνησε ήδη το 2018 και εξ αυτού 800 τόσες προτάσεις έχουν κατατεθεί. Άρα βλέπετε πόσο επιτυχημένη είναι αυτή η πρωτοβουλία ή οι πρωτοβουλίες. Είναι πολύ σημαντικό για μας να έχουμε τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου σε αυτή τη συμφωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς, λέει ο Πρόεδρος, είναι εντυπωσιακό ότι έχουν κατατεθεί πάνω από 800 προτάσεις για αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω ότι η ξηρασία είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι γειτονικέ χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωση, όπως επίσης και η επισητιστική ασφάλεια. Θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά το, χρονικό, το χρονοδιάγραμμα για αυτό το πρόγραμμα. 12 ώρα 12 Ιουλίου είναι καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών. 11 Ιουλίου, με συγχωρείτε, ψηφοφορία στην Ήτρε 3 Σεπτεμβρίου αυτού του έτους και μετά θα αποφασίσουμε για το χρονοδιάγραμμα της ε, ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελειώσαμε με αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Θα περιμένουμε λιγάκι, πολύ λίγο, γιατί έχουμε προχωρήσει πιο πολύ από ό,τι προβλεπόταν. Ο κύριος Βέστεγκαρτ, η κυρία... Α, με συγχωρείτε, πάμε στο σημείο υπερθμών 11, στην Επίτροπο. Ε, θα μας μιλήσει η κυρία Βεστάγκερ, αλλά ε, δύο λεπτά μέχρι να κάτσει. Θα διακόψουμε για δύο λεπτά. Και βλέπω έρχεται και ο κύριος Μπούζεκ, ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, έρχεται μαζί με την Επίτροπο. Good Καλό σας ε, απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε την ε, ασυνήθη τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Μαργρέτη Φεστάγκερ, Επίτροπο υπεύθυνη για θέματα ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Επίτροπε που ήρθατε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι όλοι στην Επιτροπή μας αισθανόμαστε, έχουμε μάλλον πλήρη συνέστηση, ε, ότι εκτός από την αλληλεία και την ε, γεωργία και ενδεχομένως και τις μεταφορές, ε, όλα τα άλλα στοιχεία της ε, οικονομίας μας, στην ουσία περιλαμβάνοντας θερμοδιότητες ε, της ε, Επιτροπής μας, θέματα βιομηχανίας, θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όλα πάρα πολύ σημαντικά και είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά με εσάς που είστε Επίτροπος υπεύθυνοι για θέματα ανταγωνισμού. Ήταν απόφαση των συντονιστών να σας προσκαλέσουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Το θέμα, είναι, το θέμα μας εδώ είναι ιδιαίτερος δημοφιλές. όριο ανταγωνισμού ε, στους, την εποχή του dumping και της global capacity και της παγκοσμιοποίησης. Δεν θέλουμε ακόμα να αποκαλέσουμε όλη αυτή τη διαδικασία εμπορικό πόλεμο. Ωστόσο τα πράγματα διολυσταίνουν και γίνονται επικίνδυνα και όλα αυτά έχουν επίπτωση στην έρευνα, στο εμπόριο, στις ευκαιρίες που μπορεί να έχει ε, η βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τις ευκαιρίες που μπορούν να έχουν οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Θα περιμένουμε λοιπόν κάποιες ουσιαστικές απαντήσεις ε, κυρίως προς τη βιομηχανία και προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βεβαίως θα γίνει και συζήτηση, θα λάβετε ε, ερωτήσεις, ε. αλλά πρώτα να σας ακούσουμε κυρία Επίτροπε παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ε, θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εγκάρδια λόγια που μόλις είπατε για να με καλωσορίσατε. Είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε κατάλληλο περιβάλλον ε, για τις ε, μικρές, ε, τις μεσές και τις μεγάλες επιχειρήσεις για τη βιομηχανία στην Ευρώπη, γιατί είναι αυτές που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που δημιουργούν ανάπτυξη, που δημιουργούν κέρδος εν τέλει για τους Ευρωπαίους πολίτες και την κοινωνία στο σύνολό της. Ο ανταγωνισμός βοηθάει ε, την ε, Ευρώπη έτσι ώστε να δώσει όλο της το δυναμικό. Γιατί όταν ανταγωνίζονται μεταξύ τους ε, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται τελικά να παράγουν το προϊόν το οποίο περισσότερο επιθυμούν οι καταναλωτές και με τον τρόπο αυτό αμοιβαία αναπτύσσονται. Αυτό είναι καλό για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις γιατί όταν μια εταιρεία ας πούμε ε, είναι πρωταθλήτρια στην Ευρώπη τότε μπορεί ε, να απλωθεί και να ε, κερδίσει καταναλωτές στις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται ο ανταγωνισμός και οι επιχειρήσεις γίνονται μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εμείς εγκρίνουμε ε, όλες τις συγχωνεύσεις ε, οι οποίες μας κοινοποιούνται ε, και οι οποίες δημιουργούν Ευρωπαίους πλωταθητές. Έγινε με την Peugeot, έγινε με την Opel, έγινε με την AB και με την Saab Miller ή με τη Siemens και την Καμέζα. Τα τελευταία δέκα χρόνια μελετήσαμε πάνω από 3.000 συγχωνεύσεις. 94% από αυτές τις ε, συγχωνεύσεις εγκρίθηκαν ε, χωρίς κανένα προβληματισμό όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Ε, αυτό ίσχυσε μονάχα για 6% των περιπτώσεων. Ε, και ε, στην ουσία εμείς μπλοκάραμε μονάχα 7 συγχωνεύσεις ε, πάντα τα τελευταία 10 χρόνια. Εφαρμόζουμε τους κανόνες του ανταγωνισμού σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες εμπορεύονται στην Ευρώπη σε οποιοδήποτε τομέα της βιομηχανίας και λαμβάνουμε υπόψη το κατά πόσον συμβάλλουν στην διεύρυνση του δυναμικού καινοτομίας στην Ευρώπη. Ας πούμε αναλύσαμε σε βάθος την περίπτωση της General Electric ε, όσον αφορά το αέριο και την Alstom. Ανακαλύψαμε ότι μετά από την ε, συγχώνευση ε, θα περιέκοπταν την ανάπτυξη του πιο προωθημένου, της πιο προωθημένης τουρμπίνας αερίου της Alstom και αυτού του είδους η τουρμπίνα ήταν πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε να προκύψει προκύψει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα με, χαμηλότερε με χαμηλότερες ε, εκπομπές και επομένως ε, θα βοηθούσαν ε, την επίτευξη των κλιματικών στόχων για να διατηρηθεί ο ανταγωνισμός η General Electric πούλησε ε, την επιχείρηση στην Ansaldo στην Ιταλία. Τώρα η Ansaldo έκανε επιτυχείς ε, δοκιμές μιας νέας τουρμπίνας ε, αερίου και επένδυσε σε ένα νέο εργοστάσιο το οποίο στην Ιταλία θα παράγει ακριβώς προχωρημένη τεχνολογία και που θα την πουλάει σε ολόκληρο τον κόσμο οι κανόνες που αφορούν τις ε, συγχωνεύσεις ε, υφίστανται έτσι ώστε ολόκληρη η βιομηχανία να παραμείνει σε σωστούς όρους ε, ανταγωνισμού και για κάθε βιομηχανία η οποία θέλει να προχωρήσει σε κάποια, σε συγχώνευση υπάρχουν αρκετές άλλες ευρωπαϊκές βιομηχανίες οι οποίες μπορεί να υποστούν κάποια ζημία. Οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις θέλουν να αγοράζουν ε, προϊόντα ε, και σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι επιχειρήσεις αναφέρονται σε εκατομμύρια ανθρώπους και βεβαίως κάθε βιομηχανία οπωσδήποτε θέλει να, προχωρήσει, θέλουν και οι επιχειρήσεις έναν καλό ανταγωνισμό. Ας πούμε στον τομέα του Χάλιβα χρησιμοποιείται για πάρα πολύ, μια ευρύτατη σειρά ε, προϊόντων από πλυντήρια μέχρι ε, αυτοκίνητα. Αυτό που ε, η κατασκευαστική βιομηχανία επίσης η οποία χτίζει τα σπίτια μέσα στα οποία ζούμε. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ο ανταγωνισμός να είναι σωστός έτσι ώστε οι εταιρείε οι οποίες ασχολούνται με το χάλιβα να μην αυξήσουν παράλογα τις τιμές και να έχουν καλούς όρους ανταγωνισμού. Ε, όταν ε, ε, συγχωνεύονται μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γύρονται οπωσδήποτε προβληματισμοί όσον αφορά τον ανταγωνισμό και επομένως θα πρέπει να δίνονται τα σωστά μέτρα και να, γίνει, να έχουμε τη σωστή αντιμετώπιση. Γιατί φυσικά οι εταιρείε και οι επιχειρήσεις είναι πάντα ελεύθερες να προτείνουν λύσεις έτσι ώστε να διατηρήσουν σωστό ανταγωνισμό και να μην προκαλέσουν ανησυχίες. Ε, απ' την άλλη πλευρά ε, βεβαίως ε, είναι γεγονός ότι οι εργαζόμενοι σε περίπτωση πώλησης που πρέπει, σε περίπτωση δηλαδή που πρέπει να πωληθεί κάποια, κάποιο εργοστάσιο, κάποια εγκατάσταση για να διατηρηθεί καλό επίπεδο ανταγωνισμού πάντα οι εργαζόμενοι ανησυχούν πάρα πολύ. Εμείς εμείς, ως ε, εμείς ε, ε, έχουμε κοινά συμφέροντα με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις γιατί εμείς θέλουμε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι εταιρείε αυτές. Θέλουμε να συνεχίζει ο κόσμος να αγοράζει τα προϊόντα. Θέλουμε σωστό ανταγωνισμό μέσα και από τη διαδικασία των συγχωνεύσεων και επομένω, δεν μας ενδιαφέρει να κλείνουν επιχειρήσεις και να, να, να αποκλείονται εργαζόμενοι. Ε, ε, κατά αυτή την έννοια θεωρούμε ότι έχουμε κοινούς στόχους με τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα τι σημαίνει η συγχώνευση για αυτούς. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε ε, όλες οι εμπλικόμενες επιχειρήσεις ε, να σέβονται τις εθνικές και ε, ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη διαβούλευση και την πληροφόρηση των εργαζομένων. Οι κανόνες συγχώνευσης που διέπουν τις συγχωνεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ρητά δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους και στα συνδικάτα να έρχονται σε επαφή με εμά και να λένε την άποψή τους για την συγχώνευση. Μέσα από, τη, από διαδικασίες διαβουλεύσεων η πόρτα μας θα είναι και είναι πάντοτε ανοιχτή. Αλλά φυσικά δεν είναι δυνατόν να εγκρίνουμε συγχωνεύσεις οι οποίες ε, δημιουργούν, προκαλούν ζημία στους καταναλωτές ή προκαλούν ζημία σε άλλες ε, επιχειρήσεις. Φυσικά πάντα είναι, είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση όσον αφορά ε, τους ε, κανόνες του ανταγωνισμού και για το κατά πόσον θα πρέπει περαιτέρω να προσαρμοστούν. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βελτιώνουμε διαρκώς τα πράγματα. Ε, ας πούμε ε, όσον αφορά τις ε, κρατικές επιδοτήσεις και τους κανόνες που τις διεύπουν εμείς έχουμε διευρύνει την λεγόμενη General Block Exemption αυτόν τον κανονισμό έτσι ώστε να μπορούν οι κυβερνήσεις να δίνουν κάποιες επιδοτήσεις χωρίς προηγούμενη έγκριση με την προϋπόθεση βεβαίως να ακολουθούν τους κανόνες του ανταγωνισμού. 97% των μέτρων που αφορούν κρατικές επιδοτήσεις ε, ε, ε, και επαναλαμβάνω 97% όλων των μέτρων που αφορούν επιδοτήσεις περνούν χωρίς δικιά μας διαμεσολάβηση και προχωρούν. Όταν ε, προκύπτει ζημία, ε, τότε μόνο παρεμβαίνουμε εμείς. Διαφορετικά προχωρούν ε, οι διαδικασίες. Εμείς έχουμε προτείνει επίσης το, το Ταμείο Invest της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει 15 δισεκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποστηρίξει 650 δις ευρώ επενδύσεων. Επίσης, οικοδομούν ε, ε μέσω των χρημάτων αυτών ε, και ε, τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες του μέλλοντος μέσα από εθνικά προγράμματα και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Εμείς θέλουμε μέσα από αυτά τα βήματα να κάνουμε τα πράγματα όσο γίνεται πιο εύκολα και θέλουμε η δουλειά να γίνει όσο πιο γίνεται αποτελεσματικά αλλά και εύκολα. Βεβαίως, ε, ε, βεβαίως, με όποια μέτρα και να παίρνουμε δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς και δεν είμαστε αφελείς όσον αφορά ε, την, τον συνολικό ανταγωνισμό, global competition και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Ε, οπωσδήποτε η Κίνα δυναμώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει Έχουμε επίσης τις ε, συζητήσεις ε, για τους ε, δασμούς της των Ηνωμένων Πολιτειών για τον Χάλιβα. Είναι συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Βεβαίως η Ευρώπη θα προστατέψει όσο γίνεται δυνατότερα, ισχυρότερα τα εμπορικά της ε, συμφέροντα. Ε, ο, ο γενικός ε, ισολογισμός της, εμπορικός ισολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο είναι θετικός και πιστεύουμε ότι για να έχουμε επιτυχία πρέπει να έχουμε ανοιχτές αγορές, καλό ανταγωνισμό και καινοτομία και αυτές τις αξίες θέλουμε να εξάγουμε και τον κόσμο, ε, στον κόσμο. Ε, επομένως, εμείς παίζουμε με σωστούς κανόνες ανταγωνισμούς και το, το ίδιο θέλουμε να κάνουν και οι εταίροι μας από τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε διαρκή διάλογο με την Κίνα έτσι ώστε να μειωθούν τα, ε, οι επιβλαβείς, οι επιζήμιες επιδοτήσεις. Επίσης, η Ιαπωνία θα είναι πιο ανοιχτή όσον αφορά το ίδιο θέμα και βεβαίως ε, δουλεύουμε ε, ε, στενά, σε στενή συνεργασία και με τις Ηνωμένε Πολιτείες όσον αφορά τα θέματα ανταγωνισμού. Η Ευρώπη έχει πολύ ισχυρά πόδια πάνω στα οποία να βασιστεί βγαίνοντα στον κόσμο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν απασχόληση. Είναι πολύ περισσότεροι αυτοί σε σχέση με πριν και από τις 10 ε, πιο καινοτόμες χώρες στον κόσμο, οι 10 είναι ευρωπαϊκές. Ε, ε, έχουμε λοιπόν μία όθηση την οποία θέλουμε να διατηρήσουμε και θεωρούμε ότι η Ευρώπη πραγματικά μπορεί να συνεχίσει να έχει ηγετικό ρόλο όσον αφορά τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε. Νομίζω ότι ήταν απολύτως απαραίτητο για τα μέλη της Επιτροπής μας να ακούσουν την εναρκτηρία ομιλία σας. Και ε, φυσικά υπάρχουν ε, και κάποιες ε, ερωτήσεις πολύ σημαντικές προς εσάς που αφορούν το μικρές και μεσές επιχειρήσεις και το πώς ανταγωνιζόμαστε παγκοσμίω. Θέλω να ανοίξω τώρα τη συζήτηση εκ μέρους των πολιτικών ομάδων καταρχήν για το ΕΛΚ, ο κύριος Λάγκεν. Okay, äh Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κατά τη διάρκεια της ε, θητείας σας, αναμφίβολα, πετύχατε πάρα πολλά. Η... Τα ακούτε, ακούτε τη μετάφραση, τη διερμηνία, ωραία. Οι κρατικές λοιπόν επιδοτήσεις αναμφίβολα στέφτηκαν από επιτυχία και κατά την εφαρμογή της απαγόρευσης ε, για καρτέλ. Αυτό που έχει σημασία είναι να παραμείνουν ανοιχτές οι αγορές, γιατί δεν πρόκειται μόνο για συμφωνίες για τιμές, αλλά πρόκειται κυρίως ε, για την ηλεκτρονική οικονομία να παραμείνουν ανοιχτές ε, κάποιες δίωδοι. Σήμερα μιλήσατε κυρίως για τις συγχωνεύσεις και είπατε ότι εγκρίθηκε το 94% των αιτήσεων. Σωστό. Αλλά βέβαια πολλές εξ αυτών με προαπαιτούμενα. Για μένα λοιπόν τίθεται το εξή ερώτημα. Πώς θα εξελιχθεί υπεραιτέρω το οπλοστάσιο με την έννοια ότι η αγορά σε μεγάλο βαθμό είναι παγκοσμιοποιημένη ε, τα παλιά κριτήρια στην ε, ηλεκτρονική οικονομία παίζουν ε, δευτερεύοντα ρόλο. Παράδειγμα, WhatsApp, Facebook υπήρχε ναι μεν ε, παγκοσμιοποίηση αγοράς, αλλά δεν υπήρχαν κέρδη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ήταν αρμόδια για να αξιολογεί αυτές τις συγχωνεύσεις. Τώρα, σε ένα όλο και περισσότερο παγκοσμιοποιημένο κόσμο, τι κριτήρια έχουν προκύψει και πώς θα επιτύχετε τις αλλαγές. Τι θα γίνει στο μέλλον με την πρόσβαση στις αγορές. Αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Και τρίτον, κατά την άποψή σας, τι είδους προβλήματα υπάρχουν ε, κυρίως ε, στην, στο δίκαιο που διέπει τις ε, ενισχύσεις, κυρίως προς τις επιχειρήσεις. Εκ μέρους, του SND, σοσιαλιστές, ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κυρία Επίτροπε. σας ευχαριστώ για όσα είπατε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μια περίπτωση που γνωρίζετε πολύ καλά το συλλογικό εργοστάσιο στο Γκαλάτσι. Εγώ είμαι από εκεί και από εκεί 20.000 άνθρωποι εξαρτώνται από το τι θα συμβεί με αυτό το εργοστάσιο για το αν τα παιδιά τους θα πάνε στο σχολείο και θα έχουν τι να φάνε. Πριν κάποιους μήνες ανακοινώσατε ε, το πακέτο διορθωτικών μέτρων και πήγαμε στον Καλάτσι και του εξηγήσαμε ότι εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ασχολείστε με το να υπάρχει ένας ε, μηχανισμός ε, βεβαίωσης από αυτούς που θα έρθουν να αγοράσουν το συγκρότημα στον Καλάτσι ότι θα δημιουργηθεί ένας ανταγωνιστικός πόλος για την ArcelorMittal και ότι εσείς θα παγρυπνήσετε ώστε να υπάρχει ένας μηχανισμός διαφάνειας σε ό,τι αφορά αυτό το τμήμα του πακέτου που έχει επιβληθεί στην Μιτάλη. Δυστυχώ την τελευταία περίοδο δεν έχουμε ακούσει τέτοια πράγματα ούτε ε, από εσά, ούτε από του συναδέλφου σα στην Κομισιόν. Ε, Εσεί τώρα ε, επανεπιβεβαιώνετε τη δέσμευση για τη διαφάνεια και θα υπάρχει εποπτεία αυτής της συνδιαλλαγής. Ταυτόχρονα όταν θα επιβάλλετε ε, αυτές ε, τις ε, προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι οικονομικές εγγυήσεις που θα δοθούν για όποιους θέλουν να γίνουν σοβαροί ανταγωνιστές στον τομέα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας πραγματικός ανταγωνιστής στο επίπεδο της οικονομικής συγκέντρωσης που έχει η Arsenal Mittal. Αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα της διαφάνειας ε, και της ε, δεσμεύσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένει μια ολόκληρη χώρα και απευθύνουμε μια έκκληση. Ε, πιστεύουμε ότι και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας επιβεβαιώσετε αυτό που όλοι περιμένουμε, επαγγελματισμό και διαφάνεια θα ήθελα, όπως ε, πάντα επιδεικνύεται αυτά τα στοιχεία, να μας τα δείξετε και σε αυτή την περίπτωση. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ερώτησή σας, συνάδελφε, εκ μέρου ε, των φιλελευθέρων. Η κυρία Νάχτεγκαλ. Ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Επίτροπο. Στη σημερινή κατάσταση, το Ηνωμένο Βασίλειο, ε, φυσικά, ε, μας έρθει προβλήματα με το θέμα του Brexit. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα του ανταγωνισμού. Πολλοί οικονομικοί παίκτε έχουν έδρα στο Λονδίνο και ε, φυσικά η αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ε, συρρυκνώνεται. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για τη σημερινή κατάσταση, για τον ανταγωνισμό στο χρηματοοικονομικό τομέα και τι θα μπορούσαμε ή θα πρέπει να κάνουμε τους επόμενους μήνες ως προς τον Brexit. Σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της ΓΚΟΕ, ο κύριος Γιάρο Μερικόχλητσεχ, αντιπρόεδρος. Σας ευχαριστώ, πρόεδρε. Θα μιλήσω τη γλώσσα μου, τσεχικά. Νομίζω ότι θα έχουμε τις ε, ίδιες προκλήσεις. Δηλαδή, ποιο είδος συγκέντρωση μπορούμε να επιτρέψουμε στην Ευρώπη και παγκοσμίως, πριν το χάρη σε ό,τι αφορά το γυαλί και τη συσκευασία ε, του γυαλιού, ε, έχουμε μία συγκεκριμένη συγκέντρωση. Είναι κάτι υγιές αυτό. Εγώ ε, είχα ασχοληθεί με τον τομέα του χάλιβα και ήμουν μάρτυρα της κατάρρευσης ε, του κλάδου στην Τσεχία. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω τι κάνει η Κομισιόν όταν ε, η ArcelorMittal λαμβάνει όλα τα μεγάλα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ελπίζουμε βέβαια ότι θα υπάρχει ένα θετικό αποτέλεσμα στη σημερινή δράση που έχει αναλάβει. Όμως ελπίζουμε ότι οι μεγάλες εταιρείες που συγχωνεύονται με μικρές εταιρείες ε, ουσιαστικά θα πρέπει να δούμε πώς θα δράσουν σε σχέση με τις εκπομπές, γιατί δεν υπάρχουν αυστηρά όρια για τις εκπομπές, ούτε για τα κοινωνικά ζητήματα. Οι άνθρωποι ανησυχούν τι θα τους συμβεί σε σχέση και με όσα είπε ο Ρουμάνος συνάδελφος. Και εγώ βλέπω ότι οι θέσει εργασίας απειλούνται. Παραδείγματο χάρη, ε, στην Βόρεια Γαλλία έχει τελειώσει ο τομέας του Χάλιβα στο Λουξεμβούργο συνεχίζεται, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο καιρό. Στην Τσεχική Δημοκρατία όπου εμείς στο κόμμα είχαμε μεγάλα εργοστάσια τώρα έχουμε ε, μια πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό κομμάτι στο Σάντεκαφ. Τώρα, εμένα δεν με ενδιαφέρουν μόνο οι μονομένες περιπτώσεις, αλλά όλο αυτό το θέμα είναι θέμα αρχή. Το πρόβλημα μεταξύ Ευρώπης και Κίνας βασίζεται ότι έχουμε διαφορετικά όρια, διαφορετική δυναμικότητα και για το θέμα της πρόσβασης στην αγορά. Ο ανοιχτό χαρακτήρα και η πρόσβαση θα πρέπει να διέπεται από ταυτόσιμε συνθήκε. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να έχουμε ίσου κανόνε. Έτσι λοιπόν, καταλαβαίνετε που έγκυται το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. να πούμε τώρα στους υπόλοιπους βουλευτές. Ο κύριος ε, Εντουάρ Μαρτά. Ε, Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε που είστε μαζί μας. Χαιρόμαστε που είναι εδώ. Ε, ε, φαντάζομαι ότι δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι ε, δεν συμφωνώ σε ορισμένα σημεία μαζί σας. Εγώ πιστεύω ότι οι κανόνες του ανταγωνισμού τελικά προκύπτουν από έναν κόσμο που έχει αλλάξει, που δεν είναι ο ίδιος πια. Λέτε δεν είμαστε αφελείς τότε, μα αν δεν είμαστε αφελείς είμαστε συνένοχοι. Γιατί η Κομισιόν ε, ε, αναγνωρίζει το καθεστώς αγοράς στην ε, Κίνα δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα, καταστροφικές συνέπειες, η χημεία, το, το, το χαρτί, οι σιδηρόδρομοι είναι όλοι τομείς στους οποίους η Κίνα κατέχει πάνω από 50% των συμμετοχών σε επίπεδο παγκόσμιο. Ε, ε, ε, αν προσθέσει κανείς αυτό και τις ε, πρακτικές dumping κατανοεί τι γίνεται στην αγορά και τελικά το πρώτο θύμα είναι πάντα η τιμή. Οι τιμές σε αυτές τις χώρες είναι πάντοτε τόσο χαμηλές που σίγουρα είναι εναντίον μας. Και επίσης ξεχάσατε να πείτε, δεν το αναφέρατε, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις και λόγω των κρατικών ενισχύσεων υπάρχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Ε, με όλα αυτά τα μέτρα και με όλους αυτούς τους τρόπους οπωσδήποτε η ευρωπαϊκή βιομηχανία ε, μειώνεται ε, και εν τέλει κλείνουν τα εργοστάσια. Ερωτήσεις λοιπόν. Με ποιο τρόπο λαμβάνει υπόψη η Κομισιόν το διεθνέ, τη διεθνή αγορά ως σημείο αναφοράς στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού. Δεύτερον, πώς οι αθέμητοι τρόποι ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες ανταγωνισμού. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, έχοντας σαν ε, στόχο την διατήρηση της βάσης υπολογισμού μία θέση εργασία στην βιομηχανία σημαίνει η δημιουργία τριών στους υπόλοιπους κανόνες. Με ποιο τρόπο μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό. Απαντήσατε εν μέρη, αλλά οπωσδήποτε μπορούμε να πούμε και άλλα. Τρίτον, η τεχνογνωσία μπορεί, μπορεί να θεωρηθεί σαν ε, σαν αντικειμενική αιτιολόγηση ε, και δικαιολογία των κανόνων του ανταγωνισμού. Εμείς πιστεύουμε ότι ναι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. κυρία Σπυράκη. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είναι πολύ καλό που είσαστε εδώ. Και η δική μου ερώτηση αφορά στον τομέα του χάλιβα. Στην Ελλάδα έχουμε ένα ιδιαίτερα υγιή τομέα του χάλιβα. Ε, και γι' αυτό εμείς ακολουθούμε τους κανόνες και καλούμε τους εμπορικούς μας εταίρους να πράξουν το ίδιο. Αν όμως δεν το πράξουν, θέλω να σας ε, ερωτήσω. Πιστεύετε ότι ενδέχεται να υπάρξει ένα είδος εμπορικού πολέμου και πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας και τη βιομηχανία μας βεβαίως. Η κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κυρία Βέστακα, σας καλωσορίζω. Πραγματικά είμαι ενθουσιασμένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας. Έχω τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά το μηχανισμό δυνατοτήτων, δεύτερον γενικά όσον αφορά την ανταγωνιστική πολιτική και τρίτον ερωτήματα που αφορούν στο ε, σύστημα δημόσιων ε, διαγωνισμών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέχνε έξι μηχανισμούς ε, δυνατοτήτων μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Πολωνία. Και στην ανακοίνωση τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι οι μελλοντικοί κανόνες για τον μηχανισμό δυνατοτήτων θα πρέπει να εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και θέλω να σας ερωτήσω, πριν ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό του, η, της ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί τα εγκρίνατε όλα αυτά, δεν ξέρω αν ήταν καλός ο χρονισμός. Δεύτερον, όσον αφορά τον ανταγωνισμό, το ε, έθιξαν οι συνάδελφοι, πολλοί συζητάνε για το κατά πόσον στους ε, διάφορους τομείς μπορούμε να ε, δημιουργήσουμε πρωταθλητές, παραδείγματος χάρη όπως είναι το Airbus. Έχω κατά νους του σιδηρόδρομους και τη Siemens. Το δικό σας το καθήκον ως Επίτροπος Ανταγωνισμού ε, έχετε αρμοδιότητα πέρα από τις συγχωνεύσεις ε, να στηρίζετε και μια πολιτική ανταγωνισμού προς όφελος ε, των θέσεων αγοράς. Οι ευρωπαϊκοί πρωταθλητές είναι σημαντικοί για την διεθνή αγορά. Βεβαίως και αυξάνονται οι εξαγωγικές αλλά προκύπτουν και ε, προβλήματα στην απασχόληση. Μείωση στην απασχόληση τόσο στι μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά κυρίως στους μικρούς υπεργολάβους που είναι οι πραγματικοί χαμένοι. Ρωτώ λοιπόν, αυτά στις αναλύσεις σα, πώς ακριβώς τα αξιολογείτε, με ποια κριτήρια και κατά την άποψή σα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι γενικά οι ευρωπαϊκοί πρωταθλητέ, οι European Champions, είναι καλή για την προστιθέμενη αξία και για την επαναβιομηχανοποίηση, επανεκβιομηχάνηση Τη Ευρωπαϊκή Ένωση Τώρα, ε, για του δημόσιου αγωνισμούς. Εγώ ήμουν συγκήτρια για του συνδρόμους και πέρυσι άκουσα πολλέ κραυγέ αγωνίε από ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ε, οι οποίε παραπονιούντο, παραπονούντο για ανταγωνισμό εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση και έλεγαν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ένα λοιπόν σημαντικό θέμα για να μπορεί κανεί να είναι σίγουρο ότι οι δημόσιοι διαγωνισμοί τουλάχιστον στηρίζουν την προστιθέμενη εξή στην Ευρώπη είναι ο κανονισμό του 2014. Εκεί οι ε, δημόσιοι, κατά τους δημόσιους διαγωνισμούς μπορεί να απαιτηθεί η προστιθέμενη αξία να προκύπτει στην Ευρώπη. Όμως ε, εξακολουθεί να παραμένει τζόγος ε, για τους Ευρωπαίους που καλούνται πολλές φορές να πρέπει να απορρίψουν μία προσφορά αν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει σαφής μέθοδος όσον αφορά τον καθορισμό των ποσοστών. Στην Αμερική η δημόσια η ανάθεση σε κρατικούς διαγωνισμούς, εκεί ισχύουν κάποιοι συγκεκριμένοι μαθηματικοί τύποι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια προσθήκη στην ήδη φυστάμενη οδηγία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμεί ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρος, και θα ήθελα ε, να παρακαλέσω ορισμένους αδέλφους να μην μιλάτε με αυτή την ταχύτητα γιατί μερικές φορές ξέρετε κάτι πραγματικά είναι αδύνατο να σας κατανοήσει κανείς είναι ανθρώπινα αδύνατο η κυρία Μάισνερ Λοιπόν, συνεχίζω και εγώ στα γερμανικά και θα προσπαθήσω να μιλάω σε ένα ρυθμό να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει. Έχω δύο θέματα. Ε, καταρχάς, ε, σας καλωσορίζω, κύριε Επίτροπε. Μιλήσατε για την βιομηχανία του μέλλοντος και είπατε ότι υπάρχει σκέψη για ένα σχετικό ταμείο. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν πολλές σκέψεις για την τεχνολογία και εναλλακτικέ λύσεις. Η Ευρώπη καλά τα πάει. Ε, στον ωκεανό υπάρχουν προγράμματα για τη χρήση της ενέργειας των ωκεανών. Υπάρχουν παραδείγματο παραδείγματος χάρη έπιπλα που κατασκευάζονται από, από ρήματα που έχουν ρηχθεί στους ωκεανούς. Υπάρχουν σκέψεις για εναλλακτική ενέργεια για τα σκάφη και τα πλοία. Ξέρετε όμως, σε αυτούς τους τομείς δεν δραστηριοποιούνται μόνο οι Ευρωπαίοι και οι Κινέζοι και άλλοι δεν κοιμούνται. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και τις μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά και ενδεχομένω και να λάβουν κάποια οικονομική ενίσχυση από το Ταμείο ταμείο που θέλετε να συστήσετε. Πολύ σύντομη τώρα. Είπατε με την Ιαπωνία έχουμε συμφωνία για τους ε, κανόνες ανταγωνισμού, με τις ΗΠΑ δεν έχουμε και είπατε ότι εργάζεστε για να υπάρχουν δίκαιοι ανταγωνιστικοί κανόνες με τις ΗΠΑ. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό, γιατί ξέρετε δεν είναι απλό αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ δεν είχα διερμηνία στα πολωνικά, δεν ξέρω γιατί τι έγινε. Εντάξει, καλούτσικα τα αγγλικά μου, αλλά δεν είμαι και σίγουρος ότι τα κατάλαβα όλα. Μήπως μπορείτε, υποθέτω ότι το πρόβλημα θα ήταν τεχνικής φύσεως, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Τόγια, που είναι αντιπρόεδρος τη Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πάντοτε είναι πολύ ενδιαφέρον να σα ακούμε. Θέλω να κάνω μία πολύ άμεση και σύντομη ερώτηση. Μία ερώτηση που ανέκυψε και από την κυρία Βέρνη και από τον κύριο Μαρτέν. Εσείς πολλές φορές στην παρέμβασή σας συνεχίσατε να λέτε ε, ε, περί σεβασμού του ανταγωνισμού. Ξέρουμε όλοι ότι το ε, κοινοτικό δίκαιο βασίζεται στον ανταγωνισμό και στο δίκαιο των καταναλωτών. Αλλά πού είναι η ανάπτυξη και η απασχόληση, ποια είναι δηλαδή η ισορροπία μεταξύ των δύο πυλώνων και το λέω αυτό γιατί πολλές φορές στις ομιλίες μας κάνουμε ε, ουσιαστικά μία σκέψη. Δηλαδή να σκεφτούμε ποιες αλλαγές ε, έγιναν ε, όλο το ε, δίκαιο του ανταγωνισμού πέρα από κάποιες αλλαγές γεννήθηκε σε κάποια στιγμή που οικοδομούσαμε την εσωτερική αγορά και τον εσωτερικό ανταγωνισμό. Σήμερα έχει αλλάξει ο κόσμος και ο εξωτερικός ανταγωνισμός και εμεί είμαστε ακόμη εδώ να μιλάμε για τους κανόνες του εσωτερικού ανταγωνισμού που δολοφονούν ή αποδυναμώνουν τους πρωταθλητές μας. Δεν ευνοούν λοιπόν την ανάπτυξη ούτε τη δημιουργία θέσεων που είναι κάτι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό αλλά και το δίκαιο καταναλωτών. Τι έχει κάνει η Κομισιόν ε, για να αλλάξει αυτό. Καταλαβαίνω ότι κάνετε κάποια δουλειά σε κάποια σημεία, αλλά ίσω θα πρέπει να γίνει μια βαθιά τροποποίηση, κατά την άποψή μου. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ε, έχουμε πολύ συχνά την κυρία Επίτροπο μαζί μας. Επομένως, να ακούσουμε τον κύριο Λάνγκεν για το δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πολύ σύντομη προσθήκη έχω να κάνω σε αυτό που κυβερνάει σχετικά με την οδηγία περί ανάθεση έργων και δημόσιων διαγωνισμών. Είπατε ότι η Συμφωνία Ελεύθερη μπορεί με την Ιαπωνία είναι καλή, διεκδικείται τι ίδιε συνθήκε με τι ΗΠΑ. Τώρα, υπάρχει, μία ΜΚΟ στη Γερμανία η οποία λέει ότι με αυτή τη συμφωνία με την Ιαπωνία, η Ιαπωνία είναι σε θέση να λάβει γενικά την παροχή νερού στην Ευρώπη. Ε, ρωτώ λοιπόν, εσείς την έχετε ελέγξει αυτή την οδηγία, αυτό τον κανονισμό ανταγωνισμού. Και δεύτερον, είναι αλήθεια ότι με βάση τα ισχύοντα κατακυρώνεται ο διαγωνισμός στον μειοδοτή και όχι στην καλύτερη οικονομική προσφορά. Ως εκ τούτου σημαίνει αυτό ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και τα κράτη μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στη δική τους την επικράτεια, αλλά όταν πρόκειται για ένα έργο τρίτων πρέπει να αναπευθυνθούν και σε άλλους. Και εδώ ε, στην περίπτωση της Ιαπωνίας υπάρχει κάποια εξαίρεση. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε. Έχει ανοίξει ο δεύτερος γύρος. Αν μου επιτρέπετε κύριε Επίτροπε, να προσθέσω κι εγώ κάτι. Ακούσατε κάποιες γενικές ερωτήσεις, αλλά και κάποιες πιο συγκεκριμένες. το χάρη για τη βιομηχανία του Χάλιβα. Κάποιοι συναδελφοί έθεσαν αυτό το σημαντικό θέμα. Όμως, κάθε συγκεκριμένη ερώτηση είναι σημαντική από γενική σκοπιά. Εγώ έχω μία ιδιαίτερη ερώτηση. Όμως, ε, από τη σκοπιά των παγκοσμίων ανταγωνιστών στις αγορές μας, ε, θα μπορούσε να θεωρηθεί γενική. Στι 24 Μαου, η Κομισιόν ε, υιοθέτησε μία απόφαση δέσμευση και επέβαλε στην με ένα σύνολο υποχρεώσεων για να αντιμετωπιστούν ανησυχίε ω προ τι ανταγωνιστικέ τιμέ ε, σε χώρες ριού τη Κεντρικής και Ανατολική Ευρώπης. Ε, έχουμε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστή στην ευρωπαϊκή αγορά, το ίδιο ισχύει και με την Google, στα ψηφιακά. Και σε αυτήν την περίπτωση έχουμε ένα ενεργειακό θέμα. Έχω τρεις σύντομες ερωτήσεις. Το 2013 η Κομισιόν απέριψε ε, την πρόταση της Gazprom. Θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε τις κύριες διαφορές μεταξύ εκείνων ε, των δεσμεύσεων και αυτός που δέχτηκε η Κομισιόν με την απόφαση της πριν λίγες εβδομάδες. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί αυτή η απόφαση είναι ελλειπής σε διατάξεις αποζημίωσης σε θυγόμενα μέρη, σε οκτώ κράτη-μέλη και από τις πέντε μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες στην Επιτροπή μας. Σας έστειλα μία επιστολή πριν λίγο καιρό που αφορούσε το ίδιο ζήτημα. Και αναφερόταν εκεί το εξή η έλλειψη τέτοιων μέτρων αποτελεί επικίνδυνο προηγούμενο και δεν στέλνει ένα σαφές μήνυμα για τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερασπίσει τους κανόνες της και τους πολίτες της. Και τρίτη ερώτηση το Μάρτιο η Gazprom δυστυχώς ε, αναθεώρησε υπήρξε μια αναθεώρηση στην ε, ε, υπόθεση Ναύτουγκλουμς από το δικαστήριο της Στοκόλμης. Αυτό θεωρείται ότι αποτελεί παραβίαση της απόφασης. Γιατί εμείς απογοητευτήκαμε από αυτή την απόφαση της Γκάσπρομ γιατί για μα η απόφαση περί δεσμεύσεων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. πώ θα μπορούσατε να μας εξηγήσετε τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την ερώτηση του Προέδρου. Να απαντήσω στην τρίτη ερώτηση. Η διατησία της Στοκόλμης δεν έχει επίπτωση στις τώρα δεσμευτικές δεσμεύσεις της Gazprom. Ξέρω την Gazprom ε, ε, σκέφτεται ποια βήματα νομικά θα μπορούσε να κάνει. Το παρακολουθούμε αυτό. Όμως αυτό δεν σχετίζεται με την υπόθεση Gazprom σε ό,τι αφορά το θέμα των αποζημιώσεων. Όσοι πιστεύουν ότι χρειάζονται αποζημιώσει ε, μπορούν να προσφύγουν στα εθνικά δικαστήρια. Πολύ πρόσφατα είχαμε μια πολύ σημαντική απόφαση δικαστηρίου που έλεγε ότι ανεξάρτητα από την απόφαση της Επιτροπής μπορεί να γίνει επεύθυνση στα εθνικά δικαστήρια και φυσικά ε, στη βάση αυτή μπορεί να υπάρξει και μια άποψη για το θέμα της αποζημίωσης ή μη αποζημίωσης. Νομίζω ότι ήταν ε, πολύ σημαντικό και το ότι αυτό ξεκαθαρίστηκε από τα δικαστήρια πρόσφατα. Τώρα για την πρώτη ερώτηση τι είναι σημαντικό στις ε, υποχρεωτικές ε, δεσμεύσεις ε, της Gazprom, ότι τώρα θα κάνουν μια σειρά θετικών βημάτων για την ολοκληρώση των αγορών αερίου. Αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν σε μια απόφαση απαγόρευσης δύο πράγματα. Καταρχήν, ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι, θε, ότι θα έχεις ε, το αέριό σου εκεί που θέλεις να το παραλάβεις, προκειμένου να μπορείς να το πωλήσει εκ νέου. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε έναν Πολωνό πελάτη με μια μακροπρόθεσμη σύμβαση που να θέλει να πουλήσει εκ νέου ε, το αέριο σε μία από τις χώρες της Βαλτικής. Κάποιες από αυτές τις χώρες ουσιαστικά είναι νησιά σε ό,τι αφορά την ε, το εφοδιασμό σε αέριο. Δεν υπάρχουν απαραίτητοι αγωγοί και οι δεσμεύσει που χρεώνουν την Κάσπρο να παραδώσει το αέριο ούτω ή άλλω, σαν να υπήρχε αγωγό μεταξύ του Πολωνού πελάτη στον ε, πελάτη αυτού του πελάτη. Το ίδιο ισχύει και με τη Βουλγαρία. Και αυτό θα μπορέσει να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της αγοράς αερίου. Και επίσης, είναι πιθανό σε μικροπρόθεσμα συμβάσεις ε, να υπάρχει ένα στοιχείο ε, με τις τιμές ε, καθορισμού του τιμού σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου. Βέβαια, σε αυτές τις ε, υποχρεωτικές δεσμεύσεις έχει δεχτεί η Gazprom ότι κάθε δεύτερο έτος μπορεί να ζητηθεί μία αναθεώρηση των τιμών σε περίοδο 5 ετών και το καλό είναι ότι υπάρχει ένα θετικό ε, όριο σύγκρισης ε, και είναι η τιμή στη Γερμανία και στις κάτω χώρες. Δηλαδή ακόμη και αν ανεβαίνουν όλες οι τιμές και έχουμε ε, και άνοδο των τιμών των πετρελαίων μπορεί να ζητήσεις να είναι χαμηλότερες οι τιμές γιατί μπορείς να δεις τι επικρατεί στην καθημερινή αγορά. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το τέλος της υπόθεσης Gazprom, αλλά η αρχή του η Gazprom να σέβεται πιο αυστηρούς κανόνες. Το γεγονός ότι είναι δεσμευτικές υποχρεωτικές οι δεσμεύσεις σημαίνει ότι αν τις παραβιάσουν μπορούμε να επιβάλλουμε πρόστιμο από τη στιγμή που θα δούμε ότι υπάρχει παραβίαση χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως ξέρετε καθώς ζούμε σε μια ένωση βάσει του κράτους δικαίου, χρειάζεται χρόνος και είναι σημαντικό, είναι δεσμευτικές, υποχρεωτικές αυτές οι δεσμεύσεις, ε, τις εποπτεύουμε με έναν καπιταστηματοδόχο και φυσικά ε, διασφαλίζουμε ότι τηρούνται δεσμεύσει έτσι ώστε στα θυγόμενα κράτη-μέλη οι πολίτε να έχουν ε, προσβάσιμε τιμέ για να μπορούν να παραμένουν σε ίδια επίπεδα όπως στις ε, δυτικοευρωπαϊκές χώρες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που δείξατε γενικά για τους ε, κανόνες του ανταγωνισμού. Ας δούμε λιγάκι το περιεχόμενο. Τουλάχιστον για μένα είναι σημαντικό το ότι ποτέ δεν υπήρχαν στην Ευρώπη τόσες θέσεις απασχόλησης όσες υπάρχουν σήμερα. Ποτέ η απασχόληση δεν ήταν τόσο υψηλή όσο σήμερα. Και αυτό οφείλεται και στους κανόνες ανταγωνισμού που ισχύουν σήμερα. Άρα δηλαδή τουλάχιστον γίνεται παραδεκτό ότι δεν είναι οι κανόνες ανταγωνισμού που αναχαιτίζουν την απασχόληση. Τα έλεγα μάλιστα, τολμούσα να πω ότι ισχύει σχεδόν και το αντίθετο. Γιατί αν είναι κανεί σε μια ανταγωνιστική αγορά, πρέπει κανεί να είναι προχωρημένος για να μπορεί να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Και έχετε απόλυτα δίκιο που ισχυρίζεστε ότι δεν πρόκειται για εσωτερική αγορά. Προφανώς και πρόκειται και συμφωνώ και για την παγκόσμια αγορά. Αν δείτε λιγάκι συγκεκριμένες περιπτώσει. Όταν ξεκινάμε την περίπτωση μιας συγχώνευσης, εκείνο που εξετάζουμε είναι κατά πόσον οι πελάτες ε, των υποσυγχώνευση εταιριών θα μπορούν να στραφούν σε κάποιον αργότερα. Αν δηλαδή θα αυξήσουν τις τιμές, θα περιορίσουν την επιλογή, τότε μπορεί ο πελάτης να στραφεί κάπου αλλού. Και πολύ συχνά διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες εκτός ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός κοινής αγορά που μπορεί κανείς Άρα δηλαδή τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι η αγορά αναπτύχθηκε. Και τα τελευταία χρόνια οι αγορές που είναι ενωσιακές αυξήθηκαν από 50% σε περίπου 65%. Βλέπετε λοιπόν στην ανάλυση μας ότι λαμβάνεται υπόψη το θέμα της παγκόσμιας αγοράς. Όταν προβαίνουμε στις αναλύσεις και ξεκινάμε εκ των άνω στο θέμα των περιορισμών νομίζω σε κάποιο βαθμό ισχύει το εξή. Το 94, στο 94% των ε, συγχωνεύσεων δεν υπάρχει κανένα προαπαιτούμενο. Μόνο στο 6% υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα με την έννοια ότι ανησυχούμε ε, μήπως υποφέρει ο ανταγωνισμός μετά τη συγχώνευση και ότι η εταιρεία πρέπει να βρει κάποια λύση σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το πρόβλημα, ενδεχομένως πουλώντας μια γραμμή παραγωγής μεταξύ άλλων από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει. Βεβαίως και έχουμε συζητήσει όταν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Ε, τις περιπτώσεις που είναι σαφείς, εντάξει αυτές δεν μας ενδιαφέρουν, ε, τις εξετάζουμε και ενδελεχώς αλλά ε, δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα. Ε, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε ήταν γιατί είχαμε κάποιες, κάποιους ενδιασμούς στην περίπτωση της Λουξότικα. Ανησυχήσαμε μήπως ε, υπήρχε κίνδυνος να συγχωνευτούν εταιρείε γνωστέ ε, που κατασκεύαζαν γυαλιά και τι άλλε που κατασκευάζουν σκελετό. Και απευθυνθήκαμε σε οπτικού και μα είπαν μην ανησυχείτε καθόλου. Ε, και αφού τα εξετάσαμε σε βάθο, πέρασε αυτή η γιγαντοσυχώνευση χωρί κανένα προαπαιτούμενο. Προσπαθούμε να είμαστε ε, λεπτομεριακοί και κυρίως σε περιπτώσεις όπου παίζει ρόλο το κατόφλι όταν αγοράστηκε το WhatsApp, το SOSAM και το WhatsApp και το SOSAM είναι μικρές εταιρείε ε, χωρίς συγκεκριμένο ουδό γιατί ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι γίνεται όταν συνδυάζονται και συγχωνεύονται τα δεδομένα. Ποια θα είναι μετά η θέση της εταιρεία. Λαμβάνεται και αυτό υπόψη. Κατά πόσον θα πρέπει να αλλάξουμε κάποια εργαλεία ή όχι. Ε, προφανώς αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα να το συζητήσει κανείς όταν αλλάζει η αγορά, όταν αλλάζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα, όταν αλλάζει η παραγωγή, όταν αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται η αξία. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ζήτησα από τρεις ειδικού συμβούλους να εξετάσουν ακριβώς αυτό το θέμα είναι ειδική για το δίκαιο ανταγωνισμού, για τα οικονομικά και για την τεχνολογία. Τρεις διαφορετικοί. Και αυτοί ε, θα καταθέσουν τις εκθέσεις τους ε, τον επόμενο Μάρτιο και τους ζητήσαμε και να μας συμβουλεύσουν πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Όχι μόνο αναλύσεις, αλλά και τι ακριβώς συστήνουν. Και για να τα ολοκληρώσουμε όλα αυτά, ζητήσαμε από μετόχους ε, να ασχοληθούν και αυτοί με το θέμα αυτό. Ε, έχουμε ξεκινήσει και μία ιστοσελίδα την προηγούμενη εβδομάδα, θα τρέξει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, για να μπορούν και άλλοι να τοποθετηθούν σε αυτά τα θέματα. Και πάνω σε αυτή τη βάση, ε, μέχρι στις 17 Ιανουαρίου θα έχουμε ένα μεγάλο συνέδριο ανοιχτό για να συζητήσουμε το τι ακριβώς χρειάζεται μία αγορά όπου τα μέσα παραγωγής, όπου αλλάζουν πολύ γρήγορα και τα μέσα παραγωγής και η προστιθέμενη αξία σε σχέση με την καινοτομία και αυτά γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα οποία προγραμματίζουμε είναι και τα κατάλληλα όσον αφορά το θέμα του Χαλιβουργίου στη Ρουμανία. Ξέρετε, για άλλη μια φορά θέλω να επαναλάβω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους να καταλάβουν ένα σαφές μόνιμο ότι το συμφέρον μας είναι κοινό. Για μας δεν εξυπηρετεί το να κλείσει αυτό το χαλιβουργείο γιατί αυτό το κλειστό χαλιβουργείο δεν είναι ανταγωνιστικό ο μόνος ανταγωνιστής είναι ένα ζωντανό χαλιβουργείο όπου υπάρχουν επενδύσεις στην παραγωγή αλλά και στις πωλήσει και στο να θέλει το χαλιβουργείο να είναι και σημαντικό στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν όταν μια εταιρεία προτείνει διαφοροποίηση ή έναν άλλο συνεργάτη για μας ο συνεργάτης ή ο εξαγοραστής είναι πολύ σημαντικός. Σε πάρα πολλές ε, περιπτώσεις αυτός που εξαγοράζει δεν πρέπει να έχει μόνο χρήματα αλλά και γνώση που γνωρίζει αυτό το συγκεκριμένο κλάδο γιατί είναι πολύ δύσκολο να ε, ξεκινήσει κανείς να τρέχει χωρίς καμία ανάπαυλα και να συνεχίσει η εταιρεία να δουλεύει. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ε, προσπαθούμε να έχουμε τους σωστούς αγοραστές έτσι ώστε να συνεχίσει μια εταιρεία να παραμένει ανταγωνιστική και μετά τη συγχώνευση. Και συμφωνώ όσον αφορά αυτή τη μακρά ιστορία που έχει η χαλιβουργία στην Ευρώπη. Πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Το καλό που μπορούμε να ισχυριστούμε ότι όσον αφορά τη χαλιβουργία στην Ευρώπη πράγματι εξακολουθεί να είναι ένας καλός κλάδος. Είναι ένας κλάδος ο οποίος δεν βασίζεται ε, στο να πληρώνουν οι καταναλωτές ε, τους λογαριασμούς. Γι' αυτό λοιπόν ο τομέας είναι ανταγωνιστικός και ενωτόμος ε, και με πολλούς άλλους κλάδους στην παγκόσμια αγορά. Αυτό που θέλω πραγματικά να συνεργαστούμε είναι σχετικά με τους μηχανισμούς μας ε, άμυνα στο εμπόριο, κατά του ντάμπικ, να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο ισχυροί, αν θέλουμε και αν πιστεύουμε ότι ο ανταγωνισμός είναι αθέμητος. Όπως γνωρίζετε, έχουμε 37 τέτοιες αποστολές κατά του ντάμπινγκ που τρέχουν ήδη και στο Κοινοβούλιο. Η κυρία Μάλστρομ είναι καθήλυνα αρμόδια. Ε, κάνουμε έκκληση στο Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα, βεβαίω και μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει των κανόνων του ΠΟΕ, αλλά με μεγαλύτερη ταχύτητα. Ίσως με μεγαλύτερη επιθετικότητα από ό,τι ήμασταν μέχρι τώρα, για να είμαστε και σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε σωστά. Ε, και πράγματι ελπίζω όλα αυτά θα τα περάσουμε από κοινού, γιατί είναι απαραίτητα για να πούμε και στι ευρωπαϊκέ ε, εταιρείε ότι αν έχουν πρόβλημα με αθέμητο ανταγωνισμό θα δράσουμε. Με θεμητό ανταγωνισμό βέβαια εκεί θέλουμε και εκείνε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Αλλά στον αθέμητο ανταγωνισμό θα είμαστε εκεί για να αντιμετωπίζετε Όσον αφορά το θέμα του χρηματοψηφιακού τομέα και του Brexit. Νομίζω μια τέτοια ημέρα όπως είναι η σημερινή, τι να πω κι εγώ, ανοιχτά όλα. Διότι αν υπάρχει κάποιος που, εδώ στην Άσο που ξέρει το αποτέλεσμα του Brexit, ας το πει και στους υπόλοιπους για να μπορούν και εκείνοι να προετοιμαστούν για το διακύβευμα. Προφανώς ο χρηματοψηφιακός τομέας στην Ευρώπη είναι ένα σημαντικός τομέα διότι είναι το, ένα στοιχείο τη υποδομή μα για να μπορούμε να επιτρέπουμε στι εταιρείε να δουλεύουν σωστά. Ω εκ τούτου, όλα αυτά τα παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όχι μόνο τη μεταβαστική περίοδου, αλλά και τη μελλοντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσον αφορά τώρα Ποια ήταν ακριβώς η ερώτηση? Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτησή σας. Βεβαίως, βεβαίως να την επαναλάβω. Το ένα τμήμα ήταν παρόμοιο με αυτό του συναδέλφου Μάρτεν. Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τη βιομηχανία μας από τον αθέμητο ανταγωνισμό ο οποίος αγοράζει αυτές τις μεγάλες ε, ε, επιχειρήσεις, βιομηχανίες. Η Αρσελόρ ας πούμε, έχει αγοράσει ε, τις πιο αναπτυγμένες ε, ε, χαλιβουργίες στην Ευρώπη. Και το συζητήσαμε αυτό στην Επιτροπή μας. Αυτό συνέβη και στη δικιά μου χώρα. Πώς να σας το πω. Εσείς, νομίζω, Είπατε σωστά προηγουμένως ότι ε, παρακολουθείτε ποιος θα είναι ο αγοραστής. Γιατί συμβαίνει καμιά φορά να υπάρχουν κάποιες οντότητες ε, οι οποίες δύο-τρεις μέρες πριν ας πούμε άρχισαν να λειτουργούν ε, μόλις είχαμε τέτοιο πρόβλημα στον Πόλνη γιατί καταστράφηκε η χαλιβουργία πουλήθηκε για δεύτερη φορά σε κάποιον παντελώς άγνωστο αγοραστή. Αυτή η δεύτερη ερώτηση μου λοιπόν ήταν τι γίνεται με την ε, 50% ε, αγοράστηκε από αμερικανική επιχείρηση. Εγώ ξέρω πολύ καλά τον τομέα αυτό γιατί από αυτόν προέρχομαι. Ε, στο sheet glass το ίδιο. Αγοράστηκαν τα μεγαλύτερα κομμάτια αυτής της, ε, αυτού του κλάδου. Είναι κάποιοι νέοι εισερχόμενοι, τεράστιοι και πώς μπορούμε εμείς να τους αντιμετωπίσουμε και να προστατευτούμε από αυτούς. Ε, Πρόεδρος. Είναι αδύνατο νομίζω να απαντήσει κανείς άμεσα σε αυτήν την ερώτηση αλλά είναι σημαντικό να υπάρχουν, να γίνονται τέτοιες παρατηρήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό και για να ξέρουμε πώς διαγράφεται και το μέλλον ε, των βιομηχανιών μας. Ναι. Ούτε ή άλλω καλό είναι, ε, καλό, είναι να γίνονται και τέτοιε ερωτήσει. Γιατί αν με ρωτούσετε μόνο αυτά που τα ξέρω πάρα πολύ καλά, θα ήταν πολύ σύντομη η συζήτηση. Κοιτάξτε, δεν ξέρω καθόλου, καθόλου σε καμία λεπτομέρεια ε, το θέμα της ιαλοβιομηχανίας. Ε, το σημειώνω πάντως, σημειώνω και τις πληροφορίες που μου δώσατε, να τις μελετήσω. Η δεύτερη πρόταση ενώπιον του Κοινοβουλίου που είναι σημαντική είναι η πρόταση των, ε, του ελέγχου των εμέσων επενδύσεων. Υπάρχουν πολλές τέτοιε ενδιαφέρουσε προτάσεις, αλλά το σημαντικό είναι ίσως να ξέρει κανείς ε, εάν ε, ο, γνωρίζουμε πράγματα για τον επενδυτή ή αν μπορούμε να πούμε κάτι για τον ε, επενδυτή. υπάρχουν χώρες οι οποίες ήδη προβλέπουν μηχανισμούς προστασίας. Θα μπορούσαν όλα τα κράτη να έχουν τέτοιους μηχανισμούς ελέγχου, screening mechanism, έτσι ώστε ε, να ε, ξεχωρίσουμε αυτούς τους επενδυτές οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο επενδύουν για τους σωστούς λόγους. Εγώ το προσυπογράφω αυτό, γιατί πιστεύω ότι ε, θέλουμε, ζούμε σε έναν κόσμο που ο ανταγωνισμός δεν είναι πάντα ο σωστός, που οι κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι πάντα αυτοί που θα έπρεπε να είναι και επομένως θα πρέπει να ξέρουμε, να ξέρουμε κάποια πράγματα να γίνεται έλεγχος ε, για τις άμεσες επενδύσεις, τις έμεσες, ε, τις επιδοτήσεις κλπ. Και ε, θα πρέπει να μελετούμε και να βλέπουμε εάν η επένδυση γίνεται για τους σωστούς λόγους. Και τέλος θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να μειώσουμε τις επιζήμιες επιδοτήσεις. Και βέβαια το σημαντικό είναι να κάνουμε και κάποια βήματα. Ίσως δεν έχουν λυθεί τα πάντα, αλλά ε, καλύτερα είναι να κάνουμε κάτι παρά να μην κάνουμε τίποτα. Και σε αυτό το θέμα δουλεύω πολύ κοντά ε, και αποκοινούμε την Σεσίλια. στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου δυόμιση ε, χρόνια πριν ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις σχετικά με ε, τη γεωργία. Ίσως δεν είναι σημαντικό το θέμα αυτό, δεν αφορά τη δική σας επιτροπή, αλλά ε, ήταν πραγματικά αποφάσεις ιδιαίτερα σημαντικές. Αυτό που θέλουμε είναι η δυνατότητα γρήγορης εφαρμογής μέτρων καταπολέμησης του dumping. Θέλουμε να ξέρουμε ότι οι επενδύσεις γίνονται για τους σωστούς τρόπους θέλουμε να είμαστε σε θέση να μπλοκάρουμε τις επιζήμιες ε, δημόσιες επιδοτήσεις. Και σας είπα, με την Κίνα έχει ξεκινήσει ο διάλογος, έχουμε και κάποιες συμφωνίες και με την Ιαπωνία το ίδιο. Όσον αφορά ε, τους μηχανισμούς δυνατήτων, capacity mechanism, δυναμικότητας. Θέλουμε να δημιουργήσουμε σε όλη την Ευρώπη τέτοιες ε, δυνατότητες τέτοιους μηχανισμούς ε, δυναμικότητας. Το κοινό σημείο είναι ότι τέτοιοι μηχανισμοί είναι απαραίτητοι για τα κράτη-μέλη και θα πρέπει βεβαίως ε, ε, να φαίνεται αυτό και να προκύπτει από τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, θέλουν, ε, έχουν στόχο την, ε, είναι πρόσκαιροι ε, και δεν έχουν στόχο καθόλου να διατράξουν τους όρους του ανταγωνισμού. Επομένως, ο, η νομοθεσία θα πρέπει να είναι ανάλογη έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσει να μεταρρυθμίσει την αγορά. Και η Ενεργειακή Ένωση θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη, εάν και εφόσον προκύψει κάποια ε, κάποιο πρόβλημα, να βοηθήσουν ε, η μία χώρα την άλλη. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η capacity mechanisms ε, δεν είναι μόνιμη και επίσης ε, δίνουν δυνατότητες ε, για διασυνοριακή ε, προμήθεια, καθώς επίσης λαμβάνουν υπόψη και τις ανάγκες της ζήτησης. Και υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί σύμφωνα με τους οποίους εάν από τη μία πλευρά υπάρχει ένα πικ στη ζήτηση, από την άλλη να μειώνεται ε, η κατανάλωση. Ε, ε, η νομοθεσία αλλάζει, δίνονται όμως και κάποια επιπλέον μέτρα όπως αυτό, το οποίο δεν είναι μόνιμο όπως είπα, είναι πρόσκαιρο και απλώς μπορεί να βοηθήσει σε δεδομένες στιγμές. Όσον αφορά τις δημόσιες, τους δημόσιους διαγωνισμούς, δεν το ξέρω πολύ καλά το θέμα, είναι άλλη αρμόδια επίτροπος. Έγιναν πάντως αλλαγές έτσι ώστε να μην γίνεται απλά σύγκριση τιμών, γιατί η τιμή δεν είναι το α και το ω ε, είναι ο τρόπος παραγωγής, ε, είναι το, η υπηρεσία aftermarket service ε, κλπ. Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθεια έτσι ώστε στις προκηρύξεις ακόμα να είναι σωστές οι προκηρύξεις για να πάρουν και τις σωστές προσφορές. Εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι πολύ σημαντικό να ε, να ε, χτίζονται οι υποδομές, να προχωρούν τα έργα και αυτά. Είναι θέματα πολύ πιο σημαντικά από ότι η τιμή ε, ξέρει αυτή καθεαυτή. Επίσης, ρωτήσατε ποιοι είναι οι πρωταθλητές. Εμείς δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, Ευρωπαίους πρωταθλητές. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ε, ακόμα και οι πρωταγωνιστές, ακόμα και οι πρωταθλητές, ακόμα και οι μεγάλοι αντιμετωπίζουν τους ίδιους όρους ε, ανταγωνισμού. Υπάρχουν και καλά παραδείγματα τα οποία ανέφερα πριν. Ας πούμε η Αμπέινμπεφ. Είναι από τα μεγαλύτερα ε, από τους μεγαλύτερους ομίλους μπύρας. και ε, ε, πραγματικά ε, υπήρχε λίγος ανταγωνισμός ε, στις, στον τομέα της μπύρας και τώρα οι, οι περισσότερες μπύρες είναι ευρωπαϊκές. δεν πρέπει να υπάρξει αντίφαση ανάμεσα ε, στους Ευρωπαίους πρωταθλητές ας πούμε και τον ανταγωνισμό. Ε, ε, το σημαντικό είναι όλοι να διέπονται από τους ίδιους κανόνες. Το σημαντικό είναι να παραμένεις ανταγωνιστή, ανταγωνιστικός απέναντι στους ανταγωνιστές σου, ακριβώς απέναντι σε αυτούς που είναι απέναντί σου. Τελευταία ερώτηση. Με ποιο τρόπο μπορούν να έχουν πρόσβαση ε, στα, στους ευρωπαϊκούς πόρους ε, οι μικρές επιχειρήσεις. Μαζί θα προχωρήσουμε έτσι ώστε ε, αυτό να συμβεί και εν ώψη της Ένωσης των Κεφαλαίων Συζητούμε πολύ για τις μεγάλες βιομηχανίες, για την χαλιβουργία ας πούμε, αλλά όπως είπε και ο πρόεδρος αρχικά, ε, η σπονδυλική στήλη της Ευρώπης είναι οι μικρό-μεσαίες επιχειρήσεις, είναι υπεργολάβοι, είναι αυτοί που κάνουν τη δουλειά στο τέλος. Και επομένως ε, ε, οι βιομηχανίες είναι εξίσου σημαντικές με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν για αυτές. Ευχαριστούμε πολύ. Uh, Μπορούμε να έχουμε δύο ακόμα ερωτήσει. Γιατί είναι πολύ σπάνιο να σας συναντάμε, ο κύριο Μαρτέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απλώ ε, ήθελα να τονίσω αυτό που είπε ο συνάδελφο από την ΚΟΕ. Περιμένετε, δεν τελείωσα. Αν μου δώσετε το λόγο, θα το χρησιμοποιήσω. Θα αναφερθήκατε σε ένα παράδειγμα, κυρία Βεστάγκερ. Εγώ ευχαριστούμε όταν λέτε κάθε φορά ο Ευρωπαίος καταναλωτής και στην περίπτωση της ε, χαλιβουργίας ε, στις ArcelorMittal είπατε ότι πραγματικά απευθύνθηκα σε εσά κάποιοι πελάτες ε, ότι αυτές οι δραστηριότητε ArcelorMittal θα είχαν αντίκτυπο στους τιμές. Αλλά πραγματικά ποιο μπορεί να πιστέψει αυτή την ηλικιότητα. Δηλαδή ότι η ευρωπαϊκή αγορά είναι μια κλειστή αγορά, υπάρχουν τείχοι και τίποτα δεν μπορεί να μπει. Αν ε, θεωρούμε, θεωρώ εγώ ότι είναι πολύ ακριβό το ευρωπαϊκό σίδηρο, ο ευρωπαϊκό σίδηρο, ποιο με εμποδίζει να αγοράσω από την Κίνα από άλλε χώρε. Το 2008 είχαμε 40 εκατομμύρια τόνου. Σήμερα είμαστε ελληματικοί και εισάγουμε χάλιβα από Μεξικό και Βραζιλία. Πάλι η ArcelorMittal ήταν τότε. Τότε δεν θεωρούνται δεσπόζουσα θέση και η ερώτηση που έθεσε ο συνάδελφο, η διατήρηση τη τεχνογνωσία και των θέσεων εργασία, μήπω θα μπορούσε να είναι ένα κριτήριο ευελιξία ε, στου κανόνε του ανταγωνισμού. Και η περίπτωση στον Καλάτσι είναι χαρακτηριστική. Η φόβη μου για τον Καλάτσι είναι ότι αύριο θα έρθει κάποιο να εξαγοράσει, όπω ε, έγινε με την Άλκον που αγόρασε το ευρωπαϊκό αλουμίνιο. Δεν είναι τα εργαλεία που τον ενδιαφέραν. ήταν η τεχνική, η τεχνογνωσία και το αποτέλεσμα λοιπόν ποιο είναι ότι σήμερα στην Ευρώπη δεν παράγουμε καθόλου αλουμίνιο. Όλο έχει φύγει για τον Καναδά. Αυτό φοβάμαι και για τον Καλάτσι και για την Τσεχία. Είναι θέμα τεχνογνωσίας και αν θέλετε ε, πραγματικά να ξανανοίξουν τα εργοστάσια που κλείσανε στην Τσεχία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Ρουμανία, δεν θα μπορούσαμε γιατί έχουμε χάσει τεχνογνωσία και τις ικανότητές μας. Αυτό είναι το δράμα. Σας ευχαριστούμε πολύ συνάδελφε. Λοιπόν, για να απαντηθούν τέτοιε λεπτέ και ευαίσθητε ερωτήσει δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο κύριο Λάγκε, δεν... για τον τρίτο γύρο. Όχι, δεν θέλετε για τρίτο γύρο. Τέλεια. Από τον κύριο Μαρτέν μόνο λοιπόν έχετε να απαντήσετε την ερώτηση. Νομίζω ότι έχουμε διαφορετικές ε, δεξιότητες όταν εξετάζουμε το μέλλον. Γιατί δεν συμφωνώ με την πρόγνωσή σας. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία είναι ένας ε, τομέας ε, που παράγει πολλά ε, διαφορετικά προϊόντα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους από το βασικό χάλιβα σε πάρα πολύ προηγμένα προϊόντα χάλιβα που μπορείς να βρεις στην αγορά και γι' αυτό είναι κάπως δύσκολο να αναγνωρίσω μια τόσο ομή εικόνα για το τι συμβαίνει. Δυστυχώς, εκτός αν γίνει κάτι πολύ δραματικό στην παγκοσμία οικονομία, πιστεύω ότι παγκοσμίω όταν ε, θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται με την ε, υπερβολική παραγωγή. Και στο χάλιβα έχουμε ακριβώς υπερβολική παραγωγή. Και στο φόρουμ για το Χάλιβα υπόθηκε αυτό, συμμετείχαν οι ΙΠΑ και οι Ευρωπαίοι για να το συζητήσουν αυτό το θέμα. Ο λόγος που είναι ενδιαφέρον να, να αναγνωρίσουμε τις διαφορές στα προϊόντα Χάλιβα είναι ότι ταξιδεύουν ε, πολύ διαφορετικές αποστάσεις. Για κάποια προϊόντα Χάλιβα, ναι, μπορείς να το αγοράσεις εκτός Ευρώπης γιατί ε, ο χρόνος της μεταφοράς ε, και η παράδοση έγκαιρη δεν είναι τόσο σημαντική όσο άλλα θέματα και όταν βλέπουμε αυτές τις συγχωνεύσεις ε, αναλύουμε πώς ταξιδεύει ο χάλιβας, σε ποιον στρέφονται οι άνθρωποι αν αυξηθούν οι τιμές από το συνεθή πολιτή. Και βλέπουμε διάφορα μοντέλα σε ό,τι αφορά στο χάλιβο. Ορισμένα προϊόντα δεν ταξιδεύουν και πολύ μακριά, γιατί είναι ιδιαίτερα απαραίτητα και όχι μόνο το ίδιο το προϊόν χάλιβα, αλλά και η διαπίστευση ποιότητα, η ικανότητα τη έγκαιρη παράδοση, το ε, γεγονό ότι μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο το χρειαστεί θα έχει παραπάνω από το προϊόν. Και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι στην Ευρωπαϊκή χαλιβουργία βλέπεις τα πάντα και τη γραμμή της παραγωγής από τους διάφορους τρόπους ε, ε, παραγωγής ε, ε, καθαρού κάλυφα μέχρι τα ιδιαίτερα προηγμένα προϊόντα και συγκρίνουμε κάποιες από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το χάλιβα που χρειάζεται από τις εισαγωγές γιατί δεν παράγεται εδώ και παραπονιούνται πάρα πολύ για τους μηχανισμούς εμπορικής άμυνας που θεωρούν ότι είναι ε, ουσιαστικά πάρα πολύ περιοριστικοί για αυτές. Και εγώ εκτιμώ αυτή την πολύ προηγμένη ανάλυση που γίνεται λαμβάνοντας υπόψη, όπως είπατε, ότι ε, ουσιαστικά με τις θέσεις εργασίας. Ε, στην Ευρώπη έχουμε 360.000 ε, ε, θέσεις εργασίας στο Χάλιβα, σε 23 χώρες, αλλά έχουμε 30 εκατομμύρια απασχολούμενους σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Χάλιβα. Και αυτές οι επιχειρήσεις είναι εξαρτώμενες όχι μόνο στο θέμα της ποσότητας, αλλά και για τις ανταγωνιστικές τιμές απόκτηση του προϊόντος και γι' αυτό έχουμε υποχρέωση να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα ολόκληρη της αλυσίδα αξία και όχι μόνο των ιδιαιτεροτήτων για να είμαστε σίγουροι ότι είναι ανταγωνιστικές οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Κύριε Επίτροπε. Ακόμη και αν υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ μας και δεν είμαι σίγουρη ότι εδώ είναι το τέλος της συζήτησής μας. Παρ' όλα αυτά, Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό για από τη σκοπιά τη βιομηχανία, αλλά και για το ψηφιακό τομέα, για τον ενεργειακό τομέα, ακόμη και για τη διαστημική πολιτική. Έτσι λοιπόν, η παρουσία σα ε, ως ε, Επίτροπο Παγκόσμια Αρμόδια για τον Ανταγωνισμό είναι πολύ σημαντική τώρα διάφορα θέματα, ε, αυτά δηλαδή που θίξαμε, είναι πάρα πολύ λεπτά, ευαίσθητα θέματα. Και πραγματικά θα θέλαμε να έχουμε μια ανταγωνιστική αγορά και μια ελεύθερη αγορά και φυσικά να συμμετέχουμε και στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Όπως είπατε, μπορείς μόνο αν κάποιος ανταγωνίζεται να είσαι ανταγωνιστικός. Τέλεια. Ίσως ε, αυτό είναι λοιπόν ε, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, αλλά χρειαζόμαστε και απασχόληση, θέσει εργασία. Έτσι λοιπόν ε, φαίνεται να υπάρχει βαθιά διαφωνία μεταξύ του ενό και του άλλου και από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είναι και πολύ εύκολο να προχωρήσετε. Όμω σα ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Ήταν πολύ καλή ευκαιρία για την Επιτροπή μα. Και ίσως θα έχουμε και άλλη ευκαιρία μέχρι του χρόνου το Μάρτιο ε, υπάρχουν ε, πολλές αρμοδιότητε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, και θέλουμε να, είστε, να είμαστε έτοιμοι μέχρι το χρόνο του Μάρτιο. Δεν θα είναι εύκολο. Οι διαπραγματεύσει δεν θα είναι εύκολε. Θα είναι και πρώτη φορά στην ιστορία που θα συμβεί κάτι τέτοιο. Σα ευχαριστούμε πολύ.